σε σχέση με την απαλλαγή για το 2014 που περιλαμβάνει 53 εκθέσεις από 8 εισηγητές. Η κυρία Τλαμπόβα, Σμιτ, Πίπερ, Τσαρνέτσκι, Βιστίσεν, Μακοβέη, Βόν, Μαρινέσκου. Αυτά. Επίσης θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Βίκτορ Καλντέρα που είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στη σημερινή μας συζήτηση και θα δώσω λοιπόν το λόγο στον πρώτον από τους εισηγητές μας. Για τέσσερα λεπτά η κυρία Δλαμπόβα να πάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, Πρόεδρε του Αλεκτικού Συνεδρίου, κυρίες και κύριοι. Σήμερα εγκρίνουμε ένα από τα έγγραφα κλειδί που έχουν να κάνουν με τα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Εκφράζουμε την απόψή μας, δηλαδή πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίστηκε τα κονδύλια, τα οποία είχαν να κάνουν με τις πολιτικές μας, μέσα στο οικονομικό έτος 2014. Η διαδικασία απαλλαγή είναι ένα σημείο το οποίο κάθε άνοιξη έχουμε στην ημερήσια διαταξή μας και οι συγητές υποστηρίζουν και παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους. Αυτό κάνω και εγώ σήμερα. Παρόλο που πρόκειται για μια ρουτίνα πια η διαδικασία αυτή, Θέλω να δώσω κάποιες νέες ιδέες και προτάσεις, γιατί έχουμε ένα νέο οικονομικό πλαίσιο και νέες απαιτήσεις κάτι το οποίο αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να προχωρήσουμε σε αλλαγές όσον αφορά τις προδιαγραφές ελέγχου. Και δεν πρόκειται για αυθαίρετες προτάσεις ή αλλαγές, ο σκοπός μας είναι να γίνεται καλύτερη αξιολόγηση της χρήσης των κονδυλίων, κατά πόσο δηλαδή τηρούνται οι κανόνες, αλλά και κατά πόσο οδηγούν και στα σωστά αποτελέσματα αυτά που θα θέλαμε δηλαδή και κατά πόσο τα χρήματα φτάνουν εκεί όπου τα αποτελέσματα είναι πιο απτά, που μπορούμε να βρούμε νέες προτεραιότητες και να αποφύγουμε τα στερεότυπα που ακολουθούσαμε μέχρι τώρα. Πώς μπορούμε καλύτερα να μετρήσουμε το αποτέλεσμα αυτό επίσης και να καταλήξουμε σε συμπεράσματα αφιέρωσα ολόκληρη την ε, χρονιά σε αυτές τις αλλαγές, την αλλαγή νοοτροπίας. Πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε θετικές απαντήσεις σε πολλά από τα θέματα αυτά, αν θέλουμε να παραμείνουμε αντικειμενικοί. Βέβαια, οικονομικές εξελίξεις και επενδυτικές δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζουν κάποια ανάκαμψη τελευταία, όμως οι επιπτώσεις της κρίσης εξακολουθούν να είναι Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δούμε διαφορετικά τον προπολογισμό για να αντιμετωπίσουμε ενδεχομένω νέε κρίσει. Ο ευρωπαϊκό προπολογισμό πρέπει να εξοπλίζεται με μηχανισμού ελεγκτικούς και με ελεγκτικά μέσα για να αποφεύγονται οι καταχρήσεις όταν πρόκειται για ευρωπαϊκά κονδύλια. Και να μπορεί επίση να ξέρει πώς δαπανάται κάθε ευρώ. Προσπάθεια επίσης να γίνει για τις επιδόσεις του προπολογισμού και μια πιο απλοποιημένη διαδικασία χρειάζεται. Αυτό είναι κάτι που το προτείνουν όλοι, όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και το Λεκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του του 2014. Το επιβεβαιώνουν και οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Ολλανδική Προεδρία. Συνεπώς, η απαλλαγή πρέπει να είναι ένα λογικό πολιτικό έγγραφο και όχι ad hoc μόνο να αναφέρονται διάφορα συμβάντα, θετικά ή αρνητικά που θέλουμε να συσσωρεύσουμε σε ένα κατάλογο. Προσπάθησα λοιπόν να δω πού ενδεχομένω υπάρχει λάθος διαχείριση και τη τάξη του 1% του ευρωπαϊκού ΕΠ. Προσπαθήσαμε να βρούμε λύσεις, να μην επικεντρωνόμαστε μόνο σε μερικούς τομείς. Θέλουμε να καταλήξουμε σε πολιτικούς συμβιβασμούς. Πιστεύω πάντως ότι η απαλλαγή πρέπει να είναι αντικειμενική, να έχει στέρεες βάσεις και να μην αποτελεί ένα πολιτικό εργαλείο με το οποίο να βρίσκονται σε διένεξη διάφορες χώρες μέλη μεταξύ τους. Οι διαδικασίες πιστεύω ότι μπορούν να βοηθήσουν. Είμαι πεπισμένη ότι εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν κάνει προσπάθειες να έχει έναν ευρωπαϊκό προπολογισμό ε, που να προσανατολίζεται στις επιδόσεις, τα αποτελέσματα, τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μείνει απομονωμένο. Θέλω να ευχαριστήσω τη Γραμματεία της Επιτροπής Προπολογισμών, θέλω να ευχαριστήσω επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο ε, Γιουνκέβα, και όλους τους συναδέλφους. Ευχαριστώ πολύ και παρακαλώ να είσαστε αντικειμενικοί όταν αξιολογείτε την έκθεσή μου ευχαριστούμε. επόμενο εισηγητής, η κυρία Σμιτ. Ε, Κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι εισηγήτρια για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη. και θεωρώ ότι πρέπει να καταστήσω σαφή ορισμένα σημεία. Ακόμη και φέτο. βλέπουμε τα σημεία που είχαμε αναφέρει και πέρυσι. Δηλαδή δεν έχουν αλλάξει πολλά στην αναπτυξιακή πολιτική. Είναι σημαντική είναι απαραίτητη και τη χρειαζόμαστε για να βοηθήσουμε τις χώρες της Αφρικής και να επιτρέψουμε αξιοπρεπείς συνθήκες ε, διαβίωσης στις χώρες αυτές. Αλλά λυπάμαι ότι δεν έχει αλλάξει πολύ και η κατάσταση των, προγραμμάτων, των προβλημάτων. Ο έλεγχος των ε, προγραμμάτων δεν είναι αποτελεσματικός. Πρέπει να γίνουν πολλές βελτιώσεις. Τονίζω ότι δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε υπερβολική γραφειοκρατία. Υπάρχουν επαρκή συστήματα ελέγχου ήδη, αλλά αυτό που δεν είναι επαρκές είναι ακριβώς οι μηχανισμοί να μπορούν να κάνουν τους ελέγχους, να μάθουμε από τα λάθη μας και να αντιδρούμε στις διαπιστώσεις μας. Θεωρώ ότι αυτά που είπε ο Επίτροπος Νίμιτσα ήταν πολύ σωστά. Τόνισε ότι οι πρόσφυγες που έρχονται τώρα στην Ευρώπη είναι από το Αφγανιστάν και από τη Συρία. Αυτή την, ε, σε αυτή τη συγκυρία οι ε, κάτοικοι των Αφρικανικών χωρών πηγαίνουν από τη μία στην άλλη, αλλά σύντομα μπορεί να έρθουν και σε εμά. Σε ένα κεφάλαιο λοιπόν τονίζω ότι τα μέσα του Ταμείου Ανάπτυξης πρέπει να διατίθενται με πιο ευέλικτο τρόπο. Ξέρουμε ότι έχουν μπλοκαριστεί περίπου 10 δις των πόρων χάρη σε μία έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Και ε, αυτά δεν αφορούν μόνο τα πολιετή προγράμματα, αλλά και προγράμματα τα οποία τελικά μπορεί να μην μπορέσουν να εφαρμοστούν. Το ποσό είναι περίπου ένα δις για αυτά που έχουμε χάσει. Εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την ε, κρίση των προσφύγων, τότε πρέπει να καταλάβουν και χώρες ε, που χορηγούν την αναπτυξιακή βοήθεια δεν κάνουν δώρο, είναι προσπάθεια καταπολέμησης των αιτίων ε, των μεταναστευτικών ροών. Πρέπει λοιπόν να έχουμε νέο επίπεδο η Κομισιόν μέσω της DG DEFCO και μέσω της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και, και μέσω των επιτόπου εκπροσώπων της Ένωσης που είναι ακριβώς ο συνθετικός κρίκος, όλοι αυτοί πρέπει να κάνουν περισσότερα για τα προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας. Από τα 918 προγράμματα, 428 έχουν προγράμματα εφαρμογής, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα γιατί δεν έχει έννοια να χρηματοδοτούμε προγράμματα που είναι αμφίβολης αξίας. Πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να επιτρέψουμε να γίνει επίκριση του τρόπου λειτουργίας μας και να εξαγάγουμε διδάγματα. Θα ήθελα λοιπόν τα στοιχεία αυτά ε, ε, να μην απαλληφθούν από την έκθεση. Όποιος επιτρέπει την κριτική, επιτρέπει και βελτίωση της λειτουργίας των μηχανισμών. Μέχρι το 2020 θα δώσουμε 30 δις που δεν είναι στον προπολογισμό, δηλαδή θα δοθούν απευθεία από τα Εθνικά Υπουργεία Οικονομικών προ την Κομισιόν και μετά θα πάνε στην Αφρική. Και πρέπει οπωσδήποτε ένα τέταρτο των πόρων να μπορέσουν να αξιοποιηθούν για την κρίση των προσφύγων. Και να αναφέρω και αυτά που είπε η Φεντερίκα Μογκερίνου δεν είναι δώρο αναπτυξιακή βοήθεια, είναι για μας μια αναγκαία επένδυση, μια νέα μορφή εταιρική σχέση με τους εταίρους μα στην Αφρική και να αναφέρω επίσης και τον πρόεδρο Μάρτιν Σούλτς, ο οποίος είπε το εξής. Πρέπει να βελτιωθεί η αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά να την εξαρτήσουμε με τη δημοκρατία και από το κράτος δικαίου. Δεν είναι δυνατόν κάθε δικτάτορ που καταπιέζει τον πληθυσμό του να λαμβάνει και χρηματοδότηση για να συνεχίσει να το κάνει και για να διώξει τους κατοίκους της χώρας. Είναι σαφές ότι η αναπτυξιακή βοήθεια πρέπει να αντιμετωπίσει τα αίτια των προβλημάτων και αν δεν έχουν αποτελέσματα οι ενέργειές μας να αλλάζουμε τρόπο δράσης. Δεν μπορούμε να παρατείνουμε την υπάρχουσα κατάσταση, πρέπει να αναδιαρθρώσουμε την αναπτυξιακή βοήθεια ούτω ώστε να επιδιώξουμε του καλύτερου τρόπου για να έχουμε το αποτέλεσμα επιδιώκουμε. Παρακαλώ να στηρίξετε την έκθεσή μου. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρο. Και τώρα ο κύριο Πίπα, τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ. Καταρχάς ευχαριστώ για τη συνεργασία με τους ε, σκιώδει στη διαδικασία απαλλαγή και ευχαριστώ και τους βοηθούς μας και την διοίκηση για την πληροφόρηση και τη στήριξη. Κυρίες και κύριοι, η απαλλαγή για το σώμα στο οποίο συμμετέχει κανείς είναι πάντα ευαίσθητο θέμα. Η κοινή γνώμη περιμένει να είμαστε υποδειγματικοί. Για παράδειγμα, πολιτική κτηρίων. Βεβαίω ε, είναι αναγκαίο να έχουμε περισσότερα κτίρια και το γεγονό ότι είμαστε ιδιοκτήτε μειώνει το κόστο. Αλλά ε, Θέλω να επικρίνω τον τρόπο εξυγχρονισμού των κτηρίων. Και θεωρώ ότι δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε με βέση περαιτέρω ε, επέκταση της Ένωσης. Πρέπει να βελτιώσουμε αυτά που έχουμε τώρα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε και εμείς κάποιες, ε, κάποια υποδειγματικά παραδείγματα δράσης. Το βραβείο Λουξ δεν θα πρέπει να είναι ελιτίστικο. Και πιστεύω επίσης ότι και οι ομάδε επισκεπτών πρέπει να ε, έρχονται σε εμά ε, με καλύτερη αποτελεσματικότητα, έρχονται περισσότερο με λιγότερο κόστο. Αλλά αν θέλουμε αποτελεσματικότητα πρέπει να προσαρμοζόμεθα στι νέε συνθήκε. Ενώ οι νέοι κανόνε λειτουργίας μεταξύ των τριών οργάνων μας δίνουν περισσότερη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε καλύτερα τι υπηρεσίε μα, ιδιαίτερα την επιστημονική υπηρεσία, αλλά αυτά πρέπει να, γίνει, να γίνονται χωρί ε, δέσμευση σε συγκεκριμένε ιδεολογίε να είμαστε ε, στο πνεύμα των καιρών σημαίνει ότι πρέπει να μεταρρυθμιστεί και η υπηρεσία διερμηνία και για το χρόνο εργασία και για τα τεχνικά μέσα. Δυστυχώ ε, είναι πολύ επίκαιρο και το θέμα τη ασφάλεια. Βεβαίω πρέπει να έχουμε το σωστό κόστο, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει κίνδυνο για τη λειτουργία των βουλευτών, των υπαλλήλων και των ε, επισκεπτών. Και το σωστό δεν είναι να προσπαθούμε να δώσουμε σε εξωτερικές ε, εταιρείες τέτοιες υπηρεσίες. Θα ήταν λάθος εξοικονομήσεις. Επίσης ε, έχουμε επιτύχει ορισμένα πράγματα για την εστίαση, το ε, θελούσιο ταμείο συνταξιοδότησης έχει βελτιωθεί κάπως αλλά πρέπει να γίνουν πιο γρήγορα. Θέλουμε οπωσδήποτε να έχουμε το αποτέλεσμα της εξωτερικής αξιολόγησης. Η μείωση των προνομίων και η υποδειγματική λειτουργία σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει σύγχυση μεταξύ των ε, λειτουργιών του Προέδρου και τη προεκλογική εκστρατεία. Εδώ η έκθεση επικρίνει σαφώ τον Μάρτιν Σούλτ και κάνει συστάσει και σε άλλους επικεφαλεί ψηφοδελτίων σε εκλογέ. Ο κύριο Σούλτ ορισμένε φορέ, δεν κάνει το διαχωρισμό μεταξύ των καθήκων του Προέδρου και τη ε, προσωπική του προβολή. Αυτά που κάνουν δεν είναι πάντα προ το συμφέρον συνολικά του Κοινοβουλίου και με εκπλήσει, ε, μάλλον θεωρώ ότι είναι αξιόλογο να αναφέρω, το ότι την κριτική αυτή τη συμμερίζονται και οι ε, σοσιαλιστές. Βεβαίως, σε πολλούς τομείς καταφέραμε να υπερβούμε προβλήματα του παρελθόντος. Δεν είναι δυνατόν ότι η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να περιορίζεται μόνο εδώ. Στα γραφεία μας κάνουμε όλο και περισσότερο που θα πρέπει να τα κάνει η διοίκηση κάνουμε εξοικονομίες για τον καφέ και το νερό και ορισμένοι μεταξύ μας θέλουν ε, να περιορίσουν και την δυνατότητα που έχουμε να τηλεφωνάμε και να έχουμε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Θεωρώ ότι η επιτυχία της εργασίας μας δεν έχει να κάνει μόνο με τις ε, ομιλίες ενός λεπτού. Δεν θα έπρεπε να μειώσουμε τόσο πολύ την αξιοπρέπεια της ε, δραστηριότητάς μας που να γίνουμε περίγελος. Η δουλειά μας έχει αξία και γι' αυτό δεν θα πρέπει να την υποτιμούμε. Και αυτό το αναφέρει η έκθεσή μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Για τρία λεπτά ο κύριος Τσερνιέτσκι. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, Πρόεδρε του ECA, το, πρώτο, το βασικό πρόβλημα της απαλλαγής για την Ευρώπη είναι συνεχιζόμενο εδώ και χρόνια. Πρόκειται για τη διαδικασία απαλλαγής που ξεκίνησε από τις αδυναμίες που διαπιστώθηκαν στη διάρκεια της πορείας της διαδικασίας μάλλον απαλλαγής. Θα πρέπει να δούμε τα προβλήματα που υπάρχουν και τα όσα μεταφέρονται από το 2014 στο 2015. Ιδιαίτερα Όσον αφορά το εξοπλισμούς καθώς και μεγάλες ε, μεταφορές ανάμεσα στους γραμμούς, γραμμές του προπολογισμού. Αυτά θα μπορούσαν να αποφευχθούν μέσω καλύτερου δημοσιονομικού προγραμματισμού. Οι βασικοί δείκτες θα πρέπει να αναπτυχθούν. Θα πρέπει επίσης το Συμβούλιο να ε, εγκρίνει τον κώδικα διοντολογίας που είναι απαραίτητος για τη διαφάνεια, την λογοδοσία και την ακαιρεότητα του θεσμού. Επίσης υπάρχει ανησυχητική έλλειψη διαφάνειας σε σχέση με την νομοθετική διαδικασία της διαπραγματεύσης τη θέση των κρατών μέσα στο Συμβούλιο που θα πρέπει οπωσδήποτε να αποκαλύψει τα σχετικά έγγραφα και να ε, θεσπίσει ένα σαφές πρόγραμμα σύστημα μάλλον αναφορών που θα διευκολύνει το κοινό να παρακολουθεί τις διαδικασίες αυτές με ανοιχτό και διαφανή τρόπο. Άλλο πρόβλημα είναι η έλλειψη διαφάνειας των τριμερών διαλόγων και των συνεδριάσεων διαπραγματεύσεων. Τεχνικά το Συμβούλιο θα πρέπει να αυξήσει τη διαφάνεια σε σχέση με αυτές τις διαπραγματεύσεις, λαμβάνοντας υπόψη πολιτικά προβλήματα όσον αφορά τη συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θα πρέπει να πούμε ότι το Συμβούλιο οφείλει να είναι διαφανές και ε, να λογοδοτεί στους πολίτες για τα χρήματα που του έχουν ε, εμπιστευθεί μέσω της ετήσιας ε, διαδικασίας απαλλαγής, όπως και με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Η αποτελεσματική εποπτεία τη εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού απαιτεί τη συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου μέσω μια ρύθμισης συνεργασίας. Όμως δεν υπάρχει συνεργασία ούτε και διάλογο Το Συμβούλιο δεν συμμετέχει στην διαδικασία, δεν μας δίνει τις ε, απαντήσει στι γραπτές ερωτήσεις που υποβάλλουν ή υποβάλλει η Επιτροπή ή τα μέλη της Επιτροπής μας. Το Συμβούλιο δεν συμμετέχει στις ακροάσεις ή στι συζητήσει που αφορούν τη διαδικασία δημοσιονομικού ελέγχου. Η διαδικασία της χορήγησης απαλλαγής χωριστά στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι μια παραδοσιακή πρακτική που έχει αναπτυχθεί για να εγγυηθούμε την διαφάνεια και τη δημοκρατική λογοδοσία απέναντι στους Ευρωπαίους φορολογούμενους. Τέσσερα λεπτά, Βίστησεν, επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Θέλω να σας ε, μιλήσω για την πρώτη μου έκθεση που αφορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και που στο πλαίσιο της έκθεσης ε, του ελεγκτικού συνεδρίου επέτυχε εξαιρετικά αποτελέσματα. Υπήρξαν όμως και επικρίσεις σε σχέση με το γεγονός ότι το Βέλγος, μέλος του Πρωτοδικείου, επεκρίθηκε τη διαδικασία όσον αφορά την προσθήκη δικαστών στην, στο δικαστήριο. Έπειτα υπήρξε αίτημα από πλευρά τη Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών όσον αφορά την δημοσίευση των εξωτερικών δραστηριοτήτων των δικαστών του δικαστήριου. Όσον αφορά αυτέ τι δύο πτυχέ, η ομάδα μου ανησυχεί ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, χορήγηση τη απαλλαγή προ το ελεγκτικό συνέδριο, γιατί πιστεύουμε πώ πως δημιουργήθηκε έτσι μια ε, μια ασάφεια. Τώρα, Θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου όσον αφορά την ε, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Από πολλέ απόψει ανταποκρίθηκε στα αιτήματα, στι συστάσει μάλλον που είχε υποβάλει το Κοινοβούλιο σε προηγούμενε εκθέσει. Υλοποιήθηκαν από αποταμιεύσει, εξοικονομήσει μάλλον. Συνήφθη συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και ΟΚΕ ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη λειτουργία του και άρα συστήνουμε την απαλλαγή, αν και θεωρώ πω η Επιτροπή, η ΟΚΕ, θα πρέπει μακροπρόθεσμα να εστιαστεί σε βιντεοδιασκέψεις και τη τηλεεργασία ώστε να περικόψει τις δαπάνες για οδηπορικά που είναι πολύ μεγάλες. Τώρα, όσον αφορά την απαλλαγή προς την Επιτροπή και τους διάφορους οργανισμούς και την απαλλαγή προς το Ευρωκοινοβούλιο, θα ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τη συνεργασία τους, τους οικειώδεις εισηγητές, ε, θεωρώ και θεωρούμε στην ομάδα μου ότι εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα για την απαλλαγή του Συμβουλίου, όπου δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα. Θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη προστιθέμενη εξίσου να αφορά το γενικό προϋπολογισμό για τις δράσεις που χρηματοδοτούνται κυρίως όσον αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου και την περιφερειακή ανάπτυξη. Τώρα, για τον προϋπολογισμό της Επιτροπής, θεωρούμε πως υπάρχει επικοδομητική σχέση που προκύπτει από την εργασία μας και που εκφράζει μια ολόκληρη σειρά προσδοκιών που έχουμε ήδη εκφράσει και στο παρελθόν και όσον αφορά την ανάγκη να έχουμε μεγαλύτερο όγκο πόρων, πόρων ίδιων πόρων επί τη βάση και του μεγάλου, του υψηλού μάλλον ποσοστού ε, σφάλματος είμαστε αντίθετοι για την απαλλαγή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους ε, διάφορους οργανισμούς. Τώρα, για το Ευρωκοινοβούλιο και την απαλλαγή μας δηλαδή, θεωρούμε πως θα ήταν απαραίτητο να εκφράσουμε ε, περισσότερες επικρίσεις. Είναι αλήθεια ότι υπήρξε βελτίωση στη δια... με το πέρασμα του χρόνου όσον αφορά την ε, ε, γραμματεία, αλλά όσον αφορά τον πρόεδρο Σούλτ και την δική του γραμματεία θα, είμαστε, θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο αυστηροί και όσον αφορά την εσωτερική υπηρεσία οδηγών έχουμε πρόβλημα, καθώς και με τον ε, Ευρωπαϊκό Οίκο Ιστορίας. Τώρα, για τις κοινοπραξίες, και εδώ θα καταψηφίσουμε, διότι το ποσοστό σφάλματος είναι εξαιρετικά υψηλό. Ευχαριστώ. Thank you Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος συζητητής, για 6 λεπτά η κυρία Μακοβέη. Παρακαλώ κυρία Μακοβέη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά την Επιτροπή των Περιφερειών, είμαι συγγήτρια και αποφάσισα να χορηγήσω την απαλλαγή. Και αυτό για να ενθαρρύνω την Επιτροπή των Περιφερειών, να ενθαρρύνω τις μεταρρυθμίσεις της προκειμένου να καταλάβει ότι ζούμε σε έναν κόσμο όπου κάθε ευρώ μετράει, όλες οι δαπάνες μετρούν. Πρώτη κριτική. Δεν ταξιδεύουμε με χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων. Το 2013 η Επιτροπή των Περιφερειών προέβησε 787 αποστολές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 200 ήταν στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Πάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν για τα έξοδα ταξιδιών για τους ε, τα μέλη και 4.000 για το προσωπικό. Εγώ δεν ξέρω χάρη στις αποστολές αυτές τι κέρδισαν, σίγουρα χάθηκαν όμως 9 εκατομμύρια. Τα έγγραφα που πήραμε από την Επιτροπή των Περιφερειών όσον αφορά αυτό το ζήτημα ήταν ε, εκατοντάδες σελίδες με αρκετές ασάφειες και χωρίς ακριβή νούμερα. Πρώτη κριτική λοιπόν. Όσον αφορά τα έγγραφα που πήραμε. Ζήτησα απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις σε μία σελίδα μόνο. Πήρα ως απάντηση εκατοντάδες σελίδες. Αυτό για μένα αποδεικνύει ότι δεν είναι σε θέση να θέσουν οι υπάλληλοι της Επιτροπής των Περιφερειών. Υπάρχει υπερβολική γραφειοκρατία. Το να στέλνουν εκατοντάδες σελίδες σε έναν εισηγητή ε, δείχνει αν μη τι άλλο ότι δεν μας σέβονται. Άλλη κριτική. Έγιναν προσπάθειες για να υιοθετηθούν κανόνες όσον αφορά τους whistleblowers, τους καταγγέλλοντες. εκείνοι οι οποίοι καταγγέλουν ότι δεν πάει καλά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τον Ιανουάριο του 2016 αρχίζουν να ισχύουν. Υπάρχει η περίπτωση Μακό. Είναι μια περίπτωση που επέστησε την προσοχή μας για παρατυπίες από το 2002. 13 χρόνια δηλαδή το άτομο αυτό διώκεται βρίσκεται στη δικαιοσύνη δηλαδή. Τελικά δικαιώθηκε και τον Ιούνιο η Επιτροπή των Περιφερειών θα πρέπει να έρθει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να μας πει ποια είναι η λύση. Θέλω πάντως να ευχαριστήσω τους συναδέρφους για την καλή συνεργασία που είχαμε μεταξύ μας. Πήγα στην Επιτροπή των Περιφερειών εγώ και ελπίζω να μπορέσουμε να αποφύγουμε τη γραφειοκρατία γιατί όλοι πρέπει να προσαρμοστούμε σε ένα κόσμο που αλλάζει συνεχώς. Και όσοι δεν μπορούν να προσαρμοστούν θα πρέπει να αλλάξουν δουλειά. Ήμουν επίσης συζητήτρια για την απαλλαγή όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Και δεν έχω κάποιες παρατηρήσεις. Θα έπρεπε στην ετήσια έκθεση του οργανισμού αυτό, στην ετήσια έκθεση για το 2015 δηλαδή, την επόμενη, να συμπεριλάβει κάτι για τους whistleblowers, για τους καταγγέλλοντες. Και αυτό για να τηρηθεί το καθεστώς υπαλλήλων. Επίσης, στον οργανισμό αυτό θέλω να πω ότι τα βιογραφικά των ε, ατόμων είναι δημόσια. Μπορεί κανείς να τα βρει στη Wikipedia, σε οποιαδήποτε σελίδα. Οπότε τα βιογραφικά των Ευρωπαίων ε, υπαλλήλων ε, ή άλλων δεν περιλαμβάνονται στα εμπιστευτικά έγγραφα. Η αρχή αυτή λέει ότι δεν πρέπει να δημοσιεύονται, ότι πρέπει να προστατεύονται. Όχι όμως, πρόκειται για οι υπαλλήλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση που πληρώνονται με χρήματα των φορολογούμενων και τα βιογραφικά του πρέπει να είναι γνωστά. Συστήνω λοιπόν να χορηγήσουμε την απαλλαγή πάντα για να τους ανθαρρύνουμε να προχωρήσουν σε αλλαγές. Έχω τώρα κάποια σχόλια όσον αφορά την απαλλαγή για τους οργανισμούς που έχουν να κάνουν με τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις. Ήμουνα συντάκτρια γνωμοδότησης από πλευρά της Λίμπια για τους οργανισμούς αυτούς. Πρώτα απ' όλα έχουμε ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με την δημοσίευση των βιογραφικών για πολλούς από αυτούς τους οργανισμούς. Υπάρχει ζήτημα επίσης έλλειψης προστασίας των καταγγελόντων. Και έχουμε και ένα θέμα με τη σύγκρουση συμφερόντων είναι κάτι που δεν έχει γίνει καλά κατανοητό. Δεν είναι φυσιολογικό ένας οργανισμός ο οποίος εγκρίνει, απορρίπτει ένα προϊόν, χρησιμοποιεί, απασχολεί δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι δούλευαν στην παραγωγή σε επιχειρήσεις οι οποίες παρήγαγαν μέχρι τότε το εν λόγω προϊόν. Έπειτα για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Υπάρχουν πολλές ε, δίκες, πολλές προσφυγές μάλλον, κατά του οργανισμού αυτού. πολύ έχουν ε, αναφέρει παρατυπίες. Πρέπει να προστατεύονται όσοι λένε την αλήθεια. Τέλος, για την ασφάλεια τροφίμων. Ο οργανισμός αυτός, εδώ υπάρχει μια τεράστια περίπτωση σύγκρουση συμφερόντων. Το 2016 ανακοίνωσε ο οργανισμός αυτός ότι είναι εφικτό να ορίσουν ως διευθυντή κάποιον που προέρχεται από τον κλάδο, από τη βιομηχανία τροφίμων δηλαδή. Για μας είναι απαράδεκτο αυτό. Δεν είναι δυνατόν να δίνουμε μια τέτοια θέση σε έναν τέτοιο οργανισμό, σε κάποιον ο οποίος έχει δουλέψει στο σχετικό κλάδο. Τελικά δεν ξέρουμε τι τρώμε. Και οι άνθρωποι αυτοί πλουτίζουν σε βάρος της δικιάς μας της ε, υγείας. Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε και για την Έχουμε και εκεί τέτοια φαινόμενα. Ο κύριος Βον, ευχαριστώ. Όπως και η προηγούμενη ομιλήτρια, θα χρησιμοποιήσω τώρα όλο το χρόνο ομιλίας και δεν θα επανέλθω στο τέλος της συζήτησης. Έγραψα 33 εκθέσεις για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες και φορείς. Ήταν πολλή δουλειά. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν ε, τις υπηρεσίες, το προσωπικό της ομάδας μου, τους κοιόδης, τους βοηθούς μου, τους συνεργάτες μου. Όλοι συνεργαστήκαμε. Τώρα γενικά για τη διαδικασία απαλλαγής ευχαριστώντας όλους τους συγητές των εκθέσεων απαλλαγής και, και ιδιαίτερα την εισηγήτρια για τη γενική απαλλαγή. Νομίζω ήταν θαυμάσια η έκθεσή της και πολύ αντικειμενική και νομίζω θα στηριχθεί από την πλειοψηφία του σώματος. Για τους φορείς αυτούς τους αποκεντρωμένους ευχαριστώ την Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και όλους αυτούς τους φορείς ε, που συνεργάστηκαν πολύ μαζί μου. Συνολικά οι φορείς λαμβάνουν πολλές εκθέσεις από το ελεγκτικό συνέδριο. Ήμουν σκιώδη πέρυσι για αυτές τις εκθέσεις και πρέπει να πω ότι έχει υπάρξει μεγάλη πρόοδος. Λιγότερα σχόλια από το ελεγκτικό συνέδριο και δεν υπήρχαν ε, υποπροϋποθέσεις γνώμες. Δηλαδή το συνέδριο δεν θεώρησε ότι οι λογαριασμοί δεν είναι αξιόπιστοι και δεν είχε καμία αντίρρηση για την ε, νομιμότητα και κανονικότητα των ε, ισολογισμών. Έχουν προχωρήσει λοιπόν πολλοί φορεί αυτοί στην διαδικασία εφαρμογή των ενεργειών που προέβλεπε η κοινή προσέγγιση του 2012. Υπάρχει 99% ποσοστό συμμόρφωσης και το 93% των φορέων είπαν ότι μοιράζονται υπηρεσίες με άλλους φορείς και 75% έχουν συμφωνίες συνεργασίας. Ενθαρρύνουμε λοιπόν όλους τους φορείς να εξετάσουν περαιτέρω αυτές τις δυνατότητε για να έχουμε περισσότερε εξοικονομήσει για λόγου αποτελεσματικότητα. Επιπλέον, οι φορεί έχουν τώρα και καθημερινέ γραμμέ για κοινέ διαδικασίε προμηθειών και για τη συμμετοχή στι διαδικασίε ε, προμηθειών που γίνονται από την Κομισιόν. Και αυτό θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα οι περισσότεροι φορείς. Έχουν φτάσει ήδη το στόχο τη μείωση του προσωπικού κατά 5%, αλλά ορισμένοι φορεί ανησυχούν γιατί τους έχουν ζητήσει και άλλο ένα 5% προσωπικού για ένα κοινό αριθμό ε, πόστων για αναχρησιμοποίηση. Επίσης ε, έχουμε τα απαραίτητα έγγραφα από τους ανώτερους υπαλλήλου, ε, τις δηλώσεις για μη σύγκρουση συμφερόντων και τα βιογραφικά. Ε, βεβαίως, ναι μεν πάνε καλά, οι εκθέσεις αυτές, αλλά υπάρχουν ανησυχίες και περιθώρια για βελτίωση. Για παράδειγμα, από τον Ιανουάριο το 2014, τέσσερις φορείς συνεχίζουν διαπραγματεύσεις με το κράτος μέλος ε, που τους φιλοξενεί για συμφωνίες για τα γραφεία τους. Έχει υπάρξει πρόοδος, αλλά καλό όλα τα, καλό τα κράτη-μέλη να καταλήξουν αυτές τις διαπραγματεύσεις με τους φορείς αυτούς, ούτως ώστε ε, να ε, υπάρξει συμφωνία για τα ε, γραφεία τους. Για τα υπόλοιπα προς μεταφορά πρέπει να πω ότι τα περισσότερα από αυτά τα υπόλοιπα ήταν συμφωνημένα. Αλλά υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ακυρώσεων υπολείπων. Ε, αυτό σημαίνει ότι οι πιστώσεις που μεταφέρθηκαν τελικά ήταν υπερτίμηση των αναγκών ή κατά άλλο τρόπο μη αιτιολογημένες. Χαίρομαι όμως που διαπιστώνω ότι περισσότεροι φορείς έχουν ήδη εφαρμόσει μέτρα για να αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα. Ορισμένοι φορείς αντιμετωπίζουν ακόμη πρόβλημα ισότητα ευκαιριών και εκπροσώπηση και των δύο φίλων, ιδιαίτερα σε ανώτερο επίπεδο. Ζήτησα από το δίκτυο των φορέων να μα δώσει, γιατί εμεί είμαστε η αρχή απαλλαγή, ε, μία έκθεση για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό. Επίση, καλό τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη για ισότητα των δύο φίλων όταν ορίζουν μέλη στα διοικητικά συμβούλια των φορέων. Καλό επίση του φορεί να ενισχύσουν τι προσπάθειε του για να βελτιώσουν την πολιτική δημοσίων σχέσεων, να αυξήσουν την ορατότητά του και να αυξήσουν και τη συνειδητότητα για την δραστηριότητα και τα επιτεύγματά του. Όλοι οι φορεί αυτοί κάνουν θαυμάσια δουλειά για όλου του πολίτε παντού στην Ένωση και θα πρέπει να ενημερώνουν το κοινό περισσότερο για αυτή τη δουλειά. Έτσι θα υπήρχε περισσότερη συνειδητοποίηση για τα καθήκοντά του, για το έργο του και θα ήταν καλό και για του φορεί η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού με πολύ ευρία πλειοψηφία ενέκρινε την απαλλαγή για όλους τους φορείς. Και αυτό οφειλόταν στο ότι το ελεγκτικό συνέδριο μας έδωσε μια γνωμοδότηση χωρίς επιφυλάξεις για τους οργανισμούς αυτούς και ελπίζω όταν αύριο θα ψηφίσουμε την απαλλαγή για όλους αυτούς τους οργανισμούς να χορηγήσουμε απαλλαγή σε όλους τους οργανισμούς της έκθεσής μου. Ευχαριστώ. Μαρινέσκου, τέσσερα λεπτά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, εισηγητές και τους συναδέλφους της Επιτροπής για τη συνεργασία. Υπάρχει μία μόνο τροπολογία για τις 8 εκθέσεις και φαντάζομαι πως η εργασία ε, της Επιτροπής ήταν εξαιρετική. Είναι πολύ σημαντικές οι διαδικασίε απαλλαγή. Αυτή την περίοδο μιλάμε για την οικονομική ανάπτυξη, ε, για τις δραστηριότητες της Επιτροπής και βέβαια για τις δραστηριότητες έρευνας ανάπτυξης, για την καινοτομία και για την εφαρμογή αυτών των πρακτικών ε, των αποτελεσμάτων μάλλον, των πορισμάτων στην πράξη. Πιστεύω πως ε, πλέον οι κοινέ επιχειρήσεις, οι κοινοπραξίες έχουν αποδείξει την χρησιμότητά τους για την πρακτική εφαρμογή, όπως το ΣΕΖΑΡ που έχει δείξει ήδη την, ε, την δυνατότητα εφαρμογής στα συστήματα διαχείρισης εναέρειας κυκλοφορίας είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Clean Sky έχει φτάσει αυτή η κοινή επιχείρηση σε μια φάση επίδειξης σε πολύ σημαντικών τεχνολογιών και θα μπορέσει να μας αποφέρει πολλά ωφέλη στην αεροπλοή. Ελπίζω ότι θα βρούμε τους υπόρους που χρειάζονται ώστε όλα αυτά να τεθούν και σε ε, πρακτική εφαρμογή. Τώρα, Ε, έχουμε την ε, μόνη κοινή επιχείρηση που έχει χρησιμοποιήσει, απορροφήσει μάλλον όλους τις τους πόρους για την περίοδο του, προηγούμενης, ε, του προηγούμενου πολιτικού προγράμματος, το ΙΜΗ. Τώρα, η κοινοπραξία για το ΙΤΕΡ. Το ΙΤΕΡ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και έχει αρχίσει να δείχνει ότι μπορεί να αποδώσει. Το 80% των όσων έπρεπε να γίνουν εκεί έχουν γίνει και υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την χρηματοδότηση του προγράμματος. Υπάρχει ένα σχέδιο που έχει υποβάλει ο νέος διευθυντής του ΙΤΕΡ. Αναμένουμε να εγκριθεί το σχέδιο αυτό και γι' αυτό και πρότεινα την αναβολή της απαλλαγής για το συγκεκριμένο κοινοπραξία αν και η έκθεση στηρίζει το διεθνές αυτό πρόγραμμα βεβαίως στηρίζει και την κοινοπραξία. Γνωρίζετε ότι ε, ε, έχουμε δύο ε, κοινοπραξίες, την ΕΝΕΚ και την Άρτεμις, που συγχωνεύτηκαν η κοινοπραξία Excel Artemis συνδυάστηκαν. Δεν μπορούμε να πούμε όμως κατά πόσο το, το επίπεδο σφάλματος, το περιθώριο σφάλματος ε, οφείλεται στις εθνικά στοιχεία ή όχι. Αν λοιπόν το ποσοστό σφάλματος εντάσσεται και συνδυάζεται με το επίπεδο που επιθυμούν και οι θεσμοί. Νομίζω λοιπόν ότι εφόσον υπάρχουν τα έγγραφα ε, για να μπορέσουν οι εθνικές αρχές να επαληθεύσουν θα καταλήξουμε τελικά και κατά πόσο είναι σωστά τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα. Μπορώ να χρησιμοποιήσω 6 λεπτά πρόεδρε. Έτσι δεν θα πάρω το λόγο μετά το τέλος της συζήτησης, μάλλον στο τέλος της συζήτησης. Θα ήθελα να ζητήσω για το Excel που είναι η πρώην κοινοπραξία ΕΝΙΕΚ και κοινοπραξία Άρτεμι συνδυασμένα, να ζητήσουμε λοιπόν για αυτά τα δυο αναβολή της απαλλαγής, ώστε να ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες από τις εθνικές αρχές. Τώρα, στο ψήφισμα ζητάμε από το ελεγκτικό συνέδριο να μας υποβάλει πληροφορίες λεπτομερείς σε σχέση με την αξιολόγηση των ε, συμβολών σε είδος, αλλά και γενικότερα των ιδιωτικών συμβολών. Γιατί και εκεί έχουμε ένα ποσοστό σφάλματος για το πώς εξελίσσονται οι δαπάνες σε σχέση με το ε, πολιετές ε, πρόγραμμα έρευνας, το έβδομο μάλλον πρόγραμμα έρευνας και αυτό θα πρέπει να συγκριθεί με τις ε, γραμμές του προϋπολογισμού. Ευχαριστώ λοιπόν το Ελεκτικό Συνέδριο για τη συνεργασία του. Είχαμε συνεχείς επαφές αυτή την περίοδο και ελπίζω πως θα συνεχίσουμε αυτή τη στενή συνεργασία και μέχρι το φθινόπωρο να λύσουμε αυτά τα εκρεμή προβλήματα σε σχέση με αυτές τις δύο αναβολές απαλλαγής. Ευχαριστώ. Τώρα, του Συμβουλίου. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ε, κυρία Πίτροπε, κύριοι Ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να συμμετάσχω εδώ στη συζήτηση αυτή για την χρήση προπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 στα πλαίσια της απαλλαγής 2014, έτσι όπως προβλέπεται από το άρθρο 309 της Συνθήκης. Στις 23 Φεβρουαρίου ο Υπουργό Οικονομικών Ντάσιλ Μπλουμ είχε την ε, τιμή να παρουσιάσει τις συστάσεις του Συμβουλίου όσον αφορά την ε, πρόταση για απαλλαγή. Αύριο θα ψηφίσετε. Οι πολίτες της Ευρώπης προσδοκούν από εμάς να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα των δαπανών η χρηστή οικονομική διαχείριση δεν είναι ενδιαφέρουσα μόνο για την κοινή γνώμη, είναι και νομική υποχρέωσή μας, ώστε ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός να συνάδει με τους κανόνες. Ο έλεγχος λοιπόν είναι ζωτική σημασίας. Το Συμβούλιο σύστησε η απαλλαγή αυτή να χορηγηθεί στην Επιτροπή και υπογράμμισε για ποιο λόγο πρέπει στη σύσταση αυτή. Το Συμβούλιο όμως συγχρόνως επιβεβαίωσε ότι παρόλα αυτά υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης στη χρήση του προπολογισμού. Πρώτα απ' όλα ζήτησε, ε, μάλλον ε, διαπίστωσε το Συμβούλιο ότι υπάρχει περιθώριο σφάλματος 4,4% και που πρέπει να διορθωθεί πολλές, ε, πολλοί τομείς όπως η γεωργία, η συνοχή, η έρευνα κινδυνεύουν συχνά από σφάλματα. Το Συμβούλιο εξέφρασε την ανησυχία του στο γεγονό ότι βάσει των ευρημάτων του ελεκτικού συνεδρίου, οι εθνικέ αρχέ, οι κομισιόν και ανεξάρτητοι ελεκτέ πρέπει να έχουν αρκετέ πληροφορίε για να μπορούν να εντοπίσουν και να διορθώνουν τα σφάλματα αυτά όλοι οι οικονομικοί φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων πρέπει να αναλαμβάνουν πλήρως τις ευθύνες τους και οι χώρες μέλη δηλαδή. Τώρα το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή και τις χώρες μέλη να συνεργάζονται ακόμα πιο στενά για να αποφεύγονται τα σφάλματα. Συνεπώς υπογράμμισε την ανάγκη να βελτιωθεί η ποιότητα των ελέγχων για να αποφεύγονται αλλά και να εντοπίζονται τα σφάλματα πριν κοστίσουν χρήματα στην Επιτροπή. Οπότε συμφωνώ με την κυρία Σμιτ ότι δεν χρειάζονται μόνο περισσότεροι έλεγχοι, αλλά χρειάζονται, ε, χρειάζεται εφαρμογή των ελεγκτικών μηχανισμών πρώτα απ' όλα. Κάτι το οποίο μπορεί να γίνει αποτελεσματικά, χωρίς να προσθέσουμε επίπεδα ελέγχου. Άλλη σύσταση του Συμβουλίου ήταν ότι η ανάκτηση των κονδυλίων είναι πολύ βασικό για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων. Αν υπάρχουν τέτοια σφάλματα, οι πληρωμές πρέπει να διακόπτονται μέχρι να διορθωθεί πλήρως η κατάσταση. Ποσά τα οποία έχουν πληρωθεί χωρίς να πρέπει, πρέπει να ανακτώνται χωρίς καθυστέρηση και να υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων. Το Συμβούλιο ζήτησε επίσης από την Επιτροπή να προσφέρει στην αρχή του προπολογισμού φέτος το 2016 μια πλήρη έκθεση που να περιλαμβάνει συστηματικά στοιχεία τα οποία ήδη διατίθεται στους τομείς εκείνους όπου το σφάλμα που εντοπίζεται είναι ιδιαίτερα υψηλό και να περιλαμβάνονται και αιτίε. Επίσης, το Συμβούλιο συμφωνεί με το Κοινοβούλιο ότι χρειάζεται απλοποίηση των κανόνων. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να έχουμε σωστή αξιολόγηση. Έτσι μειώνεται το διοικητικό άχθος επί των δικαιούχων και των διαφόρων αρχών, αλλά επιτρέπει επίσης πιο αποτελεσματικούς ελέγχους που θα κοστίζουν και λιγότερο. Το Συμβούλιο ε, βέβαια ευχαριστεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έργο της όσον αφορά τις υποχρεώσεις και τις πληρωμές και ζητάει συνεχή έλεγχο των ε, όσων γίνονται για να τιμήσουμε τις υποχρεώσεις μας. Ζητούμε διαφάνεια και έγκαιρη ενημέρωση όσον αφορά τις πληρωμές που γίνονται, ώστε να γίνονται καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξαν υλικά σφάλματα, παρόλα αυτά το Συμβούλιο υπογραμμίζει την ανάγκη άμβλυνσης των ε, ε, αποτελεσμάτων που έχουμε βάσει το καθάριστο εθνικού εισοδήματος. Τέλος, το Συμβούλιο ευχαριστεί για την προσέγγιση όσον αφορά τις δαπάνες και τις επιδόσεις. Το Συμβούλιο θα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τις συστάσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου να εντοπίσει το τα καλύτερα μάλλον συστήματα επιδόσεων όσον αφορά τον ευρωπαϊκό προπολογισμό σε συνεργασία με τις χώρες μέλη. Ναι, βέβαια, υπογραμμίζοντας αυτά που υπογραμμίζει και η, η συγκήτρια, ότι δηλαδή πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στις επιδόσεις. Δεν πρέπει φυσικά να προκαταλαμβάνουμε, αλλά το Συμβούλιο ευχαριστεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει. Θα υπάρξει μάλλον την προηγούμενη εβδομάδα η πρώτη συνάντηση εμπειρογνωμόνων. Είναι προφανές ότι είμαστε ακόμα μακριά από το συνολικό στόχο και γι' αυτό το Συμβούλιο θέλει κάθε χρόνο βελτίωση στα δημοσιονομικά συστήματα ώστε ο στόχος μας για μηδενικό σφάλμα να επιτευχθεί. Το Συμβούλιο συμμετέχει στις συζητήσεις για το πόσο θα βελτιωθεί η αξιολόγηση του προπολογισμού βάσει επιδόσεων. Και αυτό στα πλαίσια της μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης των επόμενων πολιτών δημοσιονομικών προοπτικών. Ζητάει το Συμβούλιο να μπορέσει και αυτό να βοηθήσει έγκαιρα. Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω. Η Προεδρία έχει αρχίσει να εργάζεται για τις επόμενες ε, πολιτικές δημοσιονομικές προοπτικές και παρακολουθεί τις συζητήσεις που γίνονται στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Το επόμενο θα είναι στις 12 Απριλίου. Στόχος είναι έγκαιρα να βρούμε δυνατότητες βελτίωσης και μεταρρυθμίσεων. Έχουν ετοπιστεί διάφορες αρχές που μπορούν να μας βοηθήσουν, να μας δείξουν τον δρόμο. Τα αποτελέσματα των συζητήσεων αυτών θα παρουσιαστούν σε μια έκθεση της Προεδρίας, στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βεβαίως και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you, Minister. And... Σας ευχαριστώ πολύ και ανακοινωνώ συναδέλφους ότι γνωρίζω πως ε, λόγω μιας ανελημμένης διοργανικής ε, δεσμεύσεως θα πρέπει να αποχωρήσετε από την Ολομέλεια, αλλά θα επανέλθετε παρακαλώ τώρα την Επίτροπο Γεωργίευα να λάβει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ αξιότιμοι εισηγητές, κύριε Υπουργέ, Πρόεδρε Καλδέρα, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ξεκινώντας, σας ευχαριστώ όλους και ιδιαίτερως τους εισηγητές που ακούσαμε να μιλούν και το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Συμβούλιο, για τη σοβαρότητα πάνω απ' όλα με την οποία προσεγγίσατε τη συζήτηση της απαλλαγής για το 2014. Είμαστε σε μια χρονική στιγμή όπου η Ευρώπη απαιτεί από εμά να επικεντρωθούμε, να αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τα κονδύλια που με θυσία ο πολίτης διαθέτει στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Έχουμε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό εφέτος την κοινή γραμμή των θεσμικών οργάνων Κοινοβουλίου, Συμβουλίου Ελεκτικού Συνεδρίου, Επιτροπής ως προς την σημασία που αποδίδουμε και την σοβαρότητα με την οποία στηριζόμαστε στον προπολογισμό. Το πόσο καλά δηλαδή αποδίδει για την ευρωπαϊκή οικονομία, για τον πολίτη, αλλά και την τήρηση των κανόνων. Ξέρω ότι μένει δουλειά να γίνει και στους δύο τομείς ακόμη. Έχουμε σταθεροποιήσει το ποσοστό του σφάλματος, πρέπει να συνεχίσουμε να το μειώνουμε και πολύ σημαντικό είναι επίσης να συνεχίσουμε να ε, αξιοποιούμε στο μέγιστο δυνατό τον προπολογισμό, να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή προσθεμένη αξία. Αναφέρθηκε νωρίτερα ότι πριν από 5-6 μέρες είχαμε την ε, συνάντηση τη διοργανική της ομάδας για τις επιδόσεις του προϋπολογισμού. Έτσι λοιπόν προσδιορίζουμε τι εννοούμε ως επιδόσεις για να συνεννοούμε σωστά πώς θα τις προσμετρούμε, πώς πιο συστηματικά θα προχωρούμε προς ε, κατάρτιση του προπολογισμού και εκτέλεσή του προσανατολισμένη προς τις επιδόσεις. Η γενική εισηγήτρια κυρία Γλαμπαγιώβα αξίζει συγχαρητηριών για την αποφασιστικότητά της να μας επιτρέψει να διευρύνουμε τις συζητήσεις μας από αυτό που αρχικά ήταν ιδιαίτερα προσανατολισμένο στην αντιμετώπιση του ποσοστού σφάλματος σε μια πολύ ξεκάθαρη ε, υπογράμμιση των αποτελεσμάτων. Τέσσερα συμπεράσματα για μας. Δεν θα είναι εξαντλητικά. Συμπληρώνω βέβαια και με αυτά που αποκόμισα από τη συζήτηση και είναι τα εξής. Καταρχάς, προς ε, ευθυγράμμιση των προτεραιοτήτων. Δεύτερον, καλύτερη ε, καταγραφή των επιδόσεων και των αποτελεσμάτων. Τρίτον, αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού σφάλματος που επεσήμανε και η κυρία Υπουργό. Και τέταρτον, αλλά πολύ σημαντικό, εξισορρόπηση μεταξύ διαχείρισης κινδύνου και αποφυγής κινδύνου. Ξεκινώ με το πρώτο σημείο λοιπόν. Καθώς προχωρούμε προς την ε, μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση, είναι η ώρα να συζητήσουμε σοβαρά και να εντοπίσουμε σε ποιο βαθμό είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε πως οι πολιτικές μας προτεραιότητες συμβαδίζουν με τον προϋπολογισμό που προβλέπουμε για αυτές. Σημασία έχει αυτό και για τα συμπεράσματα που θα ε, προκύψουν από την διάμεση αναθεώρηση των συνομικών προοπτικών, αλλά επίσης και για να μπορέσουμε να δούμε εάν αξιοποιούμε πλήρως την ευελιξία που προβλέπεται στο πολιέτε, στις πολιετές αυτές προοπτικές για τον προϋπολογισμό. Ένα άλλο κομμάτι της συζήτησης θα είναι πώς μεταφράζονται οι πολιτικοί στόχοι σε επιχειρησιακούς στόχους, κατά περίπτωση, πώς θα εξασφαλίσουμε την σωστή καταγραφή και έκθεση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται. Με τις δημοσιονομικές προοπτικές της τωρινές ξέρουμε ότι έχουμε πραγματοποιήσει ένα πολύ σημαντικό βήμα προόδου για να γίνονται σεβαστές οι προτεραιότητες και τα μέτρα υπολογισμού του τι έχουμε επιτύχει. Δεν είναι όμως όλα τέλεια. Έχουμε διδάγματα να αποκομίσουμε και ε, πάνω απ' όλα λύσεις για τις προσεχείς γενναίες προϋπολογισμών. Πάνω απ' όλα θέλω να υπογραμμίσω τον διοργανικό διάλογο και τη σημασία του, γιατί όλοι μαζί μπορούμε συνεργαζομένοι να επιτύχουμε σημαντικές ε, βελτιώσεις. Δεύτερον, χρειάζεται καλύτερη καταγραφή των επιδόσεων. Πολλές είναι οι πληροφορίες που έχουμε στη θέση μας, αλλά πρέπει να τις οργανώσουμε έτσι, ώστε να καθοδηγούν τον τρόπο με τον οποίο ορίζουμε τα κονδύλια και να ευθυγραμμιστεί έτσι η ε, καταγραφή των αποτελεσμάτων με βάση τους δείκτες μας. Εν προκειμένου, θέλω να ε, ενημερώσω ότι πρόκειται να ληφθεί μια σημαντική απόφαση εφέτος με τον συνδυασμό της έκθεσης των αποτελεσμάτων με την έκθεση του 318 της συνθήκης ε, μαζί, ώστε να έχουμε καλύτερη καταγραφή της εκτέλεσης του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Επιπλέον γνωρίζουμε πολύ καλά πως υπάρχει ανάγκη να δώσουμε κίνητρα για πρώιμη διάγνωση κινδύνων σφάλματο και σφαλμάτων, γιατί βέβαια η πρόληψη, η αποφυγή των σφαλμάτων είναι ο καλύτερος τρόπος να τα αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά μας και για την ε, πολυετή φύση των σφαλμάτων. Ξέρω ότι ε, τα ε, μετράμε σε ενιάυσια βάση, αλλά έχουν πολυετή χαρακτήρα πολλές φορές και πρέπει να δώσουμε κίνητρα για διορθώσεις, έτσι ώστε το κόστος του σφάλματος για τον πολίτη να μειωθεί. Τρίτον, εκλήθαμε να, εκλήθαμε να κοιτάξουμε με μεγαλύτερη προσοχή τα ε, μόνιμα ε, σφάλματα, τα μόνιμα ποσοστά σφαλμάτων. Θα το κοιτάξουμε και αυτό και θέλω ιδιαίτερο να υπογραμμίσω πως θα κοιτάξουμε με βάση την προηγούμενη εμπειρία από προηγούμενα πολιετή δημοσιονομικά πλαίσια, ιδιαίτερα του 2007-2013, με τους περιορισμούς βεβαίως ε, που σημαίνει το να μεταφράσουμε τους όρους του 2007-2013 σε τωρινούς όρους, ε, πρέπει να δούμε όμως ποιοι είναι οι συστημικοί κίνδυνοι και πώς μπορούμε να τους βελτιώσουμε στο μέγιστο, στο ελάχιστο. Εν τέλει, και είναι πολύ σημαντικό, θέλουμε να έχει γνώση ο καθής των δυνατοτήτων από την διαχείριση του κινδύνου. Μίλησε η Υπουργό για την απλούστευση, πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε την ευκαιρία με τις αλλαγές στο δημοσιονομικό κανονισμό να προχωρήσουμε προς την απλοποίηση. Δεν μπορούμε όμως το σφάλμα να το μηδενίσουμε, δεν μπορεί να καταστεί μηδενικό το σφάλμα και δεν μπορούμε και να αγνοήσουμε την αξιολόγηση κάποιων επιλογών που μπορεί να έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο αλλά πολύ υψηλή αξία ως δραστηριότητες. Η ανάπτυξη, Φερρυπίν. Εάν θέλουμε να αποφεύγουμε ή να αποτρέπουμε τις συγκρούσεις, να αποφεύγουμε τις καταστροφικές ε, συνέπειες της απουσίας ανάπτυξης, πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε ιδιαίτερα ε, ασταθείς συνθήκες ανάπτυξης που έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο και το ξέρουμε. Θα έχουμε τις ομάδες διαχείρισης του κινδύνου, αλλά δεν θέλουμε να τους ζητήσουμε να μην κάνουν το σωστό και να καταδικαστούν οι άνθρωποι σε, ε, στα προβλήματα αυτά λόγω της αδράνειας. Το ίδιο για τη μετανάστευση. Η ταχύτητα δράση έχει κρίσιμη σημασία και θα συνεχίσουμε να κοιτούμε με τις πολύ κρίσιμες και απαιτητικές συνθήκες όπου οι προκλήσεις ε, εντείνονται μέρα με τη μέρα και για την κυρία Κλαμπαϊόβα και την ε, παρατήρησή της με την οποία θέλω να κλείσω γιατί μας είπε ότι το, το μέλλον ε, καθίσταται παρελθόν. Θα συμπληρώσω εγώ, θα διδαχθούμε από το παρελθόν για να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον και αυτή η απαλλαγή νομίζω μας εξοπλίζει κατά τον καταλληλότερο τρόπο. Ευχαριστώ. Ε, πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Θα δώσουμε ευθύ αμέσω τον λόγο στον πρόεδρο Καλτέρη. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, κυρία Επίτροπε, Αντιπρόεδρε Γεωργέβα, κυρία Υπουργέ, το Ευρωπαϊκό Λεγνητικό Συνέδριο θεωρεί ότι είναι καλή αυτή η ευκαιρία, ούτως ώστε να συμμετάσχουμε για άλλη μια φορά στην καταληκτική τελευταία συζήτηση όσον αφορά τη δεκαετία τη απαλλαγής για την κρίση και το οικονομικό του 2014. Θα ήθελα πρώτα-πρώτα να συγχαρώ την ε, εισηγήτρια και όλους τους ε, συγκητάς που έχουν λάβει τον λόγο, αλλά ιδίως την κυρία Τιλαμπαγιώβα για το έργο το οποίο επετέλεσε. Και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου. Οι σχετικέ εκθέσει είναι πολύτιμε για τη διαδικασία την οποία τώρα ολοκληρώνουμε και ιδίω ε, η έκθεση για την ε, τον ε, προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι έτσι μπορούμε να εξαγάγουμε σημαντικά συμπεράσματα τα οποία δεν μπορούν να αγνοηθούν. Νομίζω ότι πάρα πολλά συμπεράσματα πηγάζουν από το έργο το οποίο επιτελέστη σε σχέση με αυτές τις εκθέσεις. Οπότε ε, για μας, για το, το επιτελείο μας όλα αυτά είναι πάρα πολύ ικανοποιητικά και θετικά γιατί είδαμε πόσο όσα έχουμε πει ελήφθησαν υπόψη τώρα συγκεκριμένα Όσον αφορά τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σχετική απαλλαγή, θεωρούμε ότι τώρα η πρόκληση είναι να εξασφαλιστεί ότι τα μαθήματα τα οποία αντλήθηκαν ή ε, στο παρελθόν, ιδίω ε, από την χρήση του 2014, πρόκειται να οδηγήσουν σε μακρόπνοες αλλά και ε, βραχυχρόνιες βελτιώσεις στον τρόπο χρήσης των κοινοτικών πόρων και ε, γι' αυτό σήμερα ακούσαμε για αυτού του είδους ε, την δέσμευση όλων των ε, θεσμικών οργάνων για το ότι χρειάζεται να αναλυφθεί δράση. Όμως, για να υλοποιήσουμε κάτι τέτοιο θα πρέπει αυτού του είδους τα συμπεράσματα και μαθήματα να αντικατοπτρίζονται στη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου. Επίσης και στην αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού. Και θα πρέπει αυτό να αφορά και τις τροποποίησεις όλων των αρμοδιοτήτων και λεπτομεριών όσον αφορά τις λεπτομέρειες σχετικά με τον προπολογισμό ήδη. Είπαμε από πέρσι τον Νοέμβριο αρχίσαμε ε, αυτή την καινούργια πορεία για μια νέα προσέγγιση στην ε, δαπάνη και στις επενδύσεις των κοινωνικών πόρων. Είπαμε ότι ο προπολογισμό θα πρέπει να είναι καλύτερα στοχευμένο σε σχέση με τους στρατηγικούς μας στόχους. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη ευελιξία σε καιρούς ε, ε, κρίσεως, αναφέρατε και εσείς, ε, το μεταναστευτικό. Επίσης θα πρέπει να και πιο αποτελεσματικοί σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Και βεβαίως υπάρχουν ε, ε περιθώρια για βελτίωση. όσον αφορά την ετήσια του 2014 θα πρέπει να διεκπεριώσουμε ότι εκρεμεί, θα πρέπει να μειώσουμε ε, τα λάθη σχέση με τις πληρωμές και θα πρέπει να βελτιώσουμε τις εκθέσεις όσον αφορά τα επιτευχθέντα αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θεώρησε θετικό το μήνυμα από εμάς, δέχτη τις ε, παρατηρήσεις μας, οπότε θα πρέπει όλες αυτές οι εξελίξεις να τις ε, παρακολουθήσουμε, να τις καλύψουμε με την έκθεση του 2015, την οποία τώρα προετοιμάζουμε. Φέτος ελπίζουμε ότι θα υπάρξει η δημοσιοποίηση τον Οκτώβριο νωρίτερα από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές και ευχαριστούμε την Επιτροπή και την κυρία Γεωργέβα γιατί μας βοήθησαν σε αυτή την υπόθεση αλλά βέβαια και το Κοινοβούλιο ήταν θετικό σε μια τέτοια πρόορη δημοσίευση. Θα πρέπει να ε, αναβαθμιστεί ο διάλογο με το Κοινοβούλιο και τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές ε, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα έχουμε κάποιες εκθέσεις που θα σας ε, παράσχουν ε, βοήθεια ούτως ώστε να μπορέσετε να ασκήσετε έλεγχο όσον αφορά την εκτέλεση του κοινωτικού προπολογισμού και του ευρωπαϊκού δικαίου και νομοθεσίας. Και εδώ θα καταλήξω και κυρία Πρόεδρε και βουλευτέ, λέγοντα ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αδράξει αυτή την ευκαιρία και να την αξιοποιήσει όσο γίνεται περισσότερο, τόσο ώστε ε, εκ βάθρων να αναθεωρήσει τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει η συλλογή, η δαπάνη, αλλά και η διαχείριση των ε, κοινωνικών χρημάτων για να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Πρόεδρος. Ο κύριος Πρέντα για την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών για τις απαλλαγές επ' αυτής θέλω να εκφράσω την υποστήριξή μας για τις συστάσεις που έχουν γίνει από το όργανο για τις διάφορες εκθέσεις που συζητούμε σήμερα σχετικά με τον τρόπο διαχειρίσεως του προϋπολογισμού και τις εξωτερικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν μιλούμε για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η διαχείριση των χρημάτων για στόχους εξωτερικής πολιτικής, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι τα αποτελέσματα συνεξαρτώνται και από πολλούς τοπικούς και άλλους παράγοντες. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι ο προϋπολογισμός των εξωτερικών υποθέσεων θα πρέπει να είναι πιο εύκαμπτος και πιο εύκαμπτα διαχειρίσιμος ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει καλύτερα τις ανάγκες που προκύπτουν σε ε, τρίτες χώρες και θα πρέπει να είναι και απολύτως διαφανής. Θεωρώ ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων πρέπει να μειώσουν τις καθυστερούμενες πληρωμές και πρέπει να μειώσουν τα σφάλματα βεβαίως στη χρηματοδότηση που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για εξωτερικές δράσεις. Σας ευχαριστώ. Φρουντσούλικα, η ε, Επιτροπή Αναπτύξεως. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι και αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ως εισηγητής για τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αναπτύξεως για την απαλλαγή για το Γενικό Προϋπολογισμό του 2014 και για το 8ο, 9ο, 10ο και 11ο Ευρωπαϊκά Ταμεία Αναπτύξεως έχω να εκφράσω ορισμένες ανησυχίες σχετικά με τις απαλλαγές και στην Επιτροπή Ελέγχου και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών εξεφράσαμε ανησυχίες σχετικά με τη συμπερίληψη κάποιων μη δικαιολογημένων διατυπώσεων που είχαν ληφθεί από κάποιο ανεπίσημο έγγραφο από κάποιον συνάδελφο της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού που ποτέ δεν είχαν εγκριθεί επισήμως από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Τα σημειώνω αυτά για την απαλλαγή του Ευρωπαϊκού ε, Ταμείου Αναπτύξεως και ζητεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ένα μέρος του ε, Ταμείου Περιφερειακής Αναπτύξεως για ε, θέματα μετανάστευσης. Όμως στόχος του Ταμείου Περιφερειακής Αναπτύξεως είναι να δώσει χρήματα για επενδύσεις για να μείνει ο κόσμος στον τόπο του. Σας ζητώ λοιπόν να υπερψηφίσετε τις τροπολογίες 5, 6 και 7 για να διασφαλίσετε ότι το ψήφισμα που θα ψηφιστεί αύριο αποδίδει επακριβώς τα όσα έχουν συμβεί και δεν θέτει υπό αμφισβήτηση τις θεμελιώδεις αρχές στις οποίες βασίζεται το σημαντικό αυτό ταμείο. Ευχαριστώ κύριε Κάσα. Πρόεδρε ευχαριστώ. Θέλω ιδιαίτερως ε, να αναφερθώ στις εργασίες της, των υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων η υπηρεσία για την ε, επαγγελματική κατάρτιση, για την υγεία και τα φάρμακα, πολύ σημαντικές για τις προσπάθειες που αναπτύσσουν τα κράτη, για την έρευνα, για την ανάλυση της εργασίας, για την αποφυγή κινδύνων, για την προαγωγή υγιών συνθήκων εργασίας. Ιδιαίτερα θέλουμε να εστιαστούμε στην ε, ε, εκτέλεση του προπολογισμού για τις υπηρεσίες που είναι καλή. Πρέπει να είναι χωριστές οι υπηρεσίες, πρέπει να μείνουν ε, χωριστές. Δεν πρέπει να επιβαρύνονται με υπερβολικά πολλά καθήκοντα, πρέπει χωριστά δηλαδή να εκτελούν τα καθήκοντά τους και αυτές αντίστοιχα είναι και οι συστάσεις μας για το καλό των πολιτών μας φυσικά. Ευχαριστώ, Επιτροπή των Μεταφορών και Τουρισμού, Σαλήνη. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι η απαλλαγή είναι μια ευκαιρία και όσον αφορά τις μεταφορές ούτω ώστε να προβληματιστούμε για κάτι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολλέ οι παρατηρήσει που θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά θέλω να επικεντρωθώ όσον αφορά τις επενδύσεις που είναι αποφασιστική σημασία για την πολιτική των μεταφορών νομίζω ότι βγαίνει από τη λογική της απλής πρότασης και μπαίνει στην λογική της ανάληψης δράσης γιατί έχουμε εδώ ένα ζήτημα το οποίο αφορά τις επιδόσεις τη Επιτροπής και έχουμε το πλάνο Γιούγκερ. Εμείς έχουμε επενδύσει πολλά πολιτικές απόψει εκεί πάνω γιατί έτσι ε, θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις επενδύσεις όλων των κρατών μελών. Αλλά για μας ως Επιτροπή ε, μεταφρών το μεγάλο ερωτηματικό είναι το από πού θα πάρετε αυτούς τους ε, πόρους γιατί έτσι θα βγάλετε τη, τους πόρους από εκεί που χρειάζονται ούτω ώστε να υπάρχουν οι αναγκαίοι πόροι και αναγκαίες επενδύσεις. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε από το τσεβ αυτά τα χρήματα ε, για να μπορούμε να τα κατευθύνουμε στην ίδια κατεύθυνση από, από, άλλη διάβλο. Πρόκειται για τους ιοδρόμους, οπότε παρακαλώ να μην ξαναπερικόψετε αυτούς τους πόρους, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί ε, αυτή η πάρα πολύ μεγάλη αξία του πλάνου Γιούγκερ. Η κυρία Μάλετιτς για την Περιφερειακή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Καλησπέρα κυρία Γεωργέβα. Το σφάλμα αυξήθηκε το 2014 σχέση με το 2013. Αυτό όμως δεν μας εκπλήσει. Έχουν δοθεί διαφορετικές ερμηνείες και οι ίδιοι οι οικονομικοί ελεγκτές τα έχουν μπερδέψει. Δεν ξέρουν πια τι είναι σωστό και τι είναι λάθος από αυτές τις ερμηνείες. Άρα έχουμε εδώ πληθώρα ερμηνεών και έχουμε ε, είτε πάρα πολλά τα οποία εκρεμούν και έχουμε και διάφορα, ε, διάφορα αντικανονικά ζητήματα που έχουν προκύψει. Πρόκειται για χρηματοοικονομικά μέσα που είναι τόσο περίπλοκα που το πιο εύκολο είναι παρά τα πλεονεκτήματά τους να μην τα μετέλθει, μην τα χρησιμοποιήσει κανείς. Οπότε θα πρέπει οι αντικανονικότητες να περικοπούν, να επενδύσουμε στην κατάρτιση και να αξιοποιήσουμε ε, τα μέτρα εποπτείας. Νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση και ο στόχος είναι το πώς με επιτυχία θα εφαρμόσουμε την πολιτική συνοχή και τις άλλες πολιτικές. Πρέπει να πιάσει τόπο ο προϋπολογισμός για την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της ο κύριος Ντεκάστρο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, πρώτα-πρώτα ευχαριστούμε τον εισηγητή για όλα όσα έγιναν, για το όλα σε σχέση με τη δική μας Επιτροπή. Είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία όλων των πολιτικών Το 2014 ήταν μεταβατική χρονιά για την κοινωνική πολιτική και είχαμε την, τον παλιό προγραμματισμό αλλά και εφαρμόσαμε την μεταρρύθμιση το 2015 και το 2016 είναι χρονιές όπου θα δούμε αν θα υλοποιηθούν, θα πιάσουν τόπο οι μεταρρυθμίσεις. Θα έχουμε νέους περίπλοκους κανόνες. Πρώτα-πρώτα ε, έχουμε αυτό το πρασίνισμα, το greening, που είναι η πιο σημαντική καινοτομία που εισήχθη στην ΚΑΠ. Παρ' όλα αυτά είπαμε ότι έχουμε σε σχέση με το 2013 μία μείωση των σφαλμάτων, αλλά ακόμα πρέπει να κάνουμε πολλά, ούτως ώστε να περικόψουμε την γραφειοκρατία που βαραίνει τους ε, γεωργούς. Θα πρέπει να απλουστευτεί η ΚΑΠ με εφαρμοστικές πράξεις και πράξεις κατεξιοδότηση, με ελέγχους και κυρώσεις. Άρα μεσοπρόθεσμα θα πρέπει να έχουμε την αναθεώρηση για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί όσον αφορά την δαπάνη των χρημάτων της γεωργίας και να μπορέσουμε να αυξήσουμε το όφελος για το περιβάλλον. Ο Πρόεδρος. Τουμ για την Επιτροπή Πολιτισμού. Πρόεδρε, ευχαριστώ και κάποια παρατηρήσει από την Επιτροπή Πολιτισμού. Θέλω καταρχάς να υπογραμμίσω ότι υπάρχουν κάποια σημεία από το Erasmus Plus που έχουν να κάνουν με το προηγούμενο πρόγραμμα για τη νεολαία. Λυπούμαστε που έχει διακοπεί η λειτουργία του Erasmus Plus για την Ελλάδα. Υπάρχει επίσης το θέμα της οπτικοακουστικής υπηρεσίας που επηρεάζει ε, άμεσα τις, ε, τους δικαιούχους. Δεν έχουν τηρηθεί σε πολλές περιπτώσεις οι συστάσεις ε, του ελεγκτικού συνεδρίου από σχολεία. Πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και να καλυφθούν οι θέσεις. Δεν υπάρχει αντιστοιχήση ανάμεσα στο, εφτα, στο προγραμματισμό του πολιτικού Μουσουλωμικού πλαισίου και το δεκαετή προγραμματισμό για τα θέματα της ε, παιδείας και του πολιτισμού από την Ένεση. Πρέπει επίσης να κοιτάξουμε τα θέματα της άκρας δεξιάς και των των ε, κομμάτων, ε, αλλά οι προτάσεις αυτές δεν μπορούν να γίνουν δεκτές. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω την κυρία Μακοβέη. Ας περάσουμε στον κύριο Ντυραν της Επιτροπής Συνταγματικών. Ένα λεπτό λοιπόν για να σας μιλήσω για ένα ίσον θέμα, ίσω 3 δισεκατομμύρια ευρώ όμω. Είναι αυτά που δεν μπορεί να ελέγξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 2009 και απλώ διότι Συμβούλιο και Επιτροπή παίζουν ένα είδος πινκ-πονγκ. Το Συμβούλιο αρνείται να ανοίξει του λογαριασμού του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ΔΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνείται να ενσωματώσει στους λογαριασμού τη το προπολογισμό του Συμβουλίου. Βρισκόμαστε λοιπόν σε αδυναμία Εμεί, οι κοινοβουλευτικοί να ελέγξουμε του λογαριασμούς αυτούς και ωστόσο σε ένα χρονικό σημείο που η διαφάνεια καθίσταται απόλυτα αναγκαία. Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων λοιπόν με την ευκαιρία της παρουσίας στο ημικύκλιο και των τριών θεσμικών οργάνων ζητεί να σταματήσει η κατάσταση αυτή που είναι απολύτως γελία στο νομικό επίπεδο και σκανδαλώδης στο οικονομικό. Δηλαδή ότι οι λογαριασμοί του Συμβουλίου εκφεύγουν παντός κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ευχαριστώ. Αιάλα Σέντερ, Επιτροπή Μεταφορών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πρώτα πρώτα τον ε, κύριο Καλτέρα γιατί πάντοτε η ετήσια έκθεση είναι πολύ χρήσιμη μαζί με τις επιμέρους εκθέσεις για αυτή τη φορά μας ανησυχεί το τι γίνεται ε, με το ότι το ε, λάθος του 2014 αυξήθηκε και ξέρουμε ότι τώρα για, το Ταμείο Συνοχής είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε είπαμε ότι θα πρέπει να γίνει κάποια έρευνα και δεν είναι δυνατόν να καταργηθούν οι εκ των προτέρων έλεγχοι σαν μέτρο απλούστευσης. Το είπαμε και με τον Επίτροπο κ. Μέδας και είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον. Επίσης ευχαριστούμε την ε, εισηγήτρια γιατί έτσι ε, εξαντλητικά εξήτασε ό,τι γίνεται όσον αφορά τους ελέγχους και ε, αυτό το λάβουμε υπόψη για τους μέλλοντες προϋπολογισμούς και άρα ε, για, για άλλη μια φορά μας έχει βοηθήσει η συνάδελφος επίσης και ο συνάδελφος Πίπερ ε, νομίζω ότι συνέχεια βελτιώνει τις επιδόσεις του Κοινοβουλίου τώρα που το Κοινοβούλιο προσπαθεί να ανακτήσει τον ρόλο του ως ελεγκτού και συνομοθέτη και βέβαια είμαστε κατά των μικροκομματικών επιθέσεων κατά του Πρόεδρου του Κοινοβουλίου. Επίση, το πιο σημαντικό είναι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τον Πρόεδρο γιατί προσπαθεί του να σεβαστούν το Κοινοβούλιο και κρατών και κυβερνήσεων. Ο κύριος Φέρμπερ, ευχαριστώ στην Επιτροπή Οικονομικών ασχοληθήκαμε ιδίω με, την εποπτική, με τις ε, τρεις εποπτείες ε, τραπεζών, αξιογράφων και το καθεξής. Και χαιρόμαστε που κατέληξε σε θετική γνώμη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι δηλαδή τα χρήματα δαπανήθηκαν με ορθό τρόπο. Και αυτό μας ικανοποιεί. Από την άλλη μεριά έχουμε και μια σειρά αποκριτικές σε ό,τι αφορά την μεθοδολογία των εποπτικών αυτών αρχών. Θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό το ότι μία από τις αρχές αυτές δεν κατόρθωσε να κάνει την ε, ε, πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ηλεκτρονική της τεχνολογία με τέτοιο τρόπο που να ικανοποιεί την νομοθεσία. Έχουμε λοιπόν τώρα ανάγκη ενός έτους αναστολής. Για άλλη υποπτική αρχή φαίνεται να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, δηλαδή γενικούς κανόνες, απομακρυσμένες από την ε, πραγματική νομοθεσία, παρεμβαίνοντας έτσι στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτά τα πράγματα τα σημειώνουμε στην έκθεσή μας. Ελπίζουμε ότι η απαλλαγή δεν θα, αποτελέσει συγγνώμη, μια τυπική απλά διαδικασία, αλλά θα επιτρέψει στις τρεις αυτές εποπτικές αρχές να διορθωθούν. Τότε η δική μας Επιτροπή θα είναι πραγματικά πανευτυχής. Το όνομα της Επιτροπής Αλίας, ο κ. Πλάν Πολόπης. η, το Ελληνικό Συνέδριο ε, υπέβαλε εκείνη την έκθεση που είναι ε, τέλεια και οπότε είπαμε ότι ε, το 2014 είχαμε πάρα πολύ καλές επιδόσεις το ίδιο και όσον αφορά την μεταρρύθμιση της αληθικής πολιτικής. Έχουν πάρα πολύ λίγα λάθη. Είπαμε για περικοπή προσωπικού και για πάγμα του προϋπολογισμού. Και εμείς θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να κάνουμε εξοικονομήσεις ούτω ώστε να μπορεί η, υπηρεσία σχετική να βοηθήσει για τα ό,τι αρμοδιότητες έχει στα πλαίσια της κοινή ελευθερικής πολιτικής. Και τώρα, εκ μέρους των ε, πολιτικών ομάδων, οι αγορητές, 1,5 λεπτό κύριος Τσέλερ. Ο κύριος Τσέλερ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει στην διαδικασία του προπολογισμού. Αυτό σημαίνει όμω ότι οφείλουμε να προσέχουμε ω ευρωβουλευτέ ότι τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού προϋπολογισμού χρησιμοποιούνται ορθά. Αυτό γίνεται μέσα στο shared management, δηλαδή σε κοινή διαχείριση, γιατί οι δαπάνες εκτελούνται τελικώς από τις χώρες μέλη. Να μην διστάζουμε λοιπόν να σημειώνουμε τα σφάλματα και τις ε, παρατυπίες που σημειώνονται στις χώρες μέλη όπου σημειώνονται, ώστε ο έλεγχος και η λειτουργία εποπτείας να βελτιωθούν στις χώρες αυτές. Εφόσον έχουμε ένα στόχο τη τάξη του 2% σφάλματος για την διάθεση των πιστώσεων, δεν μπορούμε να συγχωρούμε όταν το ελεγκτικό συνέδριο διαπιστώνει ότι το ποσοστό σφάλματος βρίσκεται συνεχώ πάνω από το όριο αυτό και μάλιστα πάντοτε στι ίδιε χώρε. Όταν πρόκειται για δημοσιονομικές διορθώσεις ή για την ανάκτηση χρημάτων για ορισμένες χώρες αυτό είναι πάνω από το τριπλάσιο του μέσου όρου, πρόκειται για αριθμό που υποδηλεί ότι ο προϋπολογισμός δεν εκτελέστηκε με ορθό τρόπο. Οι δε ανακτήσεις που συνεπάγεται αυτό μέσα στα πλαίσια δηλαδή των δημοσιονομικών διορθώσεων είναι χρήματα τα οποία τελικώς δεν καταλήγουν στους στόχους που είχαν θεσπιστεί, που μπορεί να είναι η εκπαίδευση, η απασχόληση κλπ. Πάντως, είναι σωστά τα εργαλεία των διορθώσεων και της ανακτήσεως των πιστώσεων, γιατί αυτά αποτελούν και την προστατευτική ασπίδα του προϋπολογισμού και επομένως του φορολογουμένου στην Ένωση. Εκ μέρους της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο κύριος Πυρήνη και δύο λεπτά. Χωρίς μικρόφωνο. Πρόεδρε. Κύριε Γεωργίευα, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να επισημάνω τρεις σκέψεις. Πρώτον, είναι πολύ σημαντικό να μας απασχολήσει ο τρόπος με τον οποίο διατίθεται χρησιμοποιείται το χρήμα του Ευρωπαίου φορολογουμένου. Αυτό το καταδεικνύει το ποστό του σφάλματος. Άρα το ποστό του σφάλματος θα είναι κύριος δείκτης για τις δραστηριότητες της Επιτροπής σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Ταυτόχρονα όμως θέλει ο πολίτης να γνωρίζει και πώς βελτιώνονται χάρη στον προϋπολογισμό οι δικές τους προοπτικές. Φερρυπίν, εάν υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για απασχόληση εάν οι δραστηριότητες που χρηματοδοτεί ο Ευρωπαϊκός Προπολογισμός ε, και εκτελεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αποβαίνουν ισοφελώς τους. Η έκθεση λοιπόν της συναδέλφου, της κυρίας Τλαμπάλοβα, είναι πολύ σημαντική διότι ε, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις πτυχές αυτές για την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της Επιτροπής. Ευχαριστώ την κυρία Σλαπάγιοβα ως συντάκτης ταυτόχρονα. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο στην έκθεση, στο σημείο 73, λέγεται ότι ο Ευρωπαίος πολίτης δεν αντιλαμβάνεται τι σημαίνει ποστό σφάλματος. Και γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελεκτικό Συνέδριο πρέπει να συνεργαστούν στενά για τον προσδιορισμό μιας μεθοδολογίας που θα προσδιορίζει το ποσοστό του σφάλματος. Χρειάζονται επίσης κοινέ μέθοδοι καταγραφής της εκτέλεσης έτσι ώστε να γνωρίζουμε πιο καλά ποιος ε, χρησιμοποιεί τα χρήματα με ποιον τρόπο. Ευχαριστώ. Κουσμουκ. Συντηρητική μεταρρυθμιστές. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Πρόεδρε του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Λαμβάνοντας το λόγο για, τον, για την εκτέλεση του προπολογισμού του 2013, θα ήθελα να αφαιρθώ στο τμήμα 3 για τις υπηρεσίες, πολύ μεγάλο και σημαντικό τμήμα του προπολογισμού. Σε σχέση με τις δαπάνες αυτές, λοιπόν, έχω να επισημάνω τα εξή σημαντικά προβλήματα. Πρώτον, το πολύ ψηλό ποσοστό σφάλματος, που σε σχέση με τις πληρωμές ανέρχεται στο 4,4% αντίστοιχο με τα έτη 2012 και 2013. Στη συνοχή και τη γεωργία 70% των συνολικών μας δαπανών το ποσοστό του σφάλματος ήταν ακόμα πιο υψηλό, 5,7% και 6,2% αντίστοιχα. το ποστό σφάλματο βέβαια δεν σημαίνει πάντοτε παρατυπίε, δεν, σημαίνει, σημαίνει πάντοτε ότι ε, πηγαίνουν χαμένα τα χρήματα, διασπαθίζονται. Μπορεί να υπάρχουν απλώ ε, νομικοί λόγοι πίσω από αυτό. Αλλά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συνεχίζεται το ποστό του σφάλματο. Επίση, έχουμε σε πολλά προγράμματα μηδενική απορρόφηση για το 2014 στο πολιτές νομικό πλαίσιο 2014-2020 λόγω καθυστέρησης της έγκρισης του κανονισμού από την Επιτροπή έχουμε μηθενική απορρόφηση και μπορεί να συνεχιστεί και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τλαμπάλοβα, φιλελεύθερη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, ομιλώ ως κοιόδηση συγγήτρια για την έκθεση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αναπτύξεως. Ευχαριστώ όλους τους κοιόδης εισηγητές καθώς και τον κύριο εισηγητή για την συνεργασία. Πολλά σημαντικά νέα στοιχεία περιλήφθηκαν στην έκθεση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αναπτύξεως για το 2013, το οποίο έχει γίνει πλέον αναπόσπαστο τμήμα όλων των κειμένων περί απαλλαγής με την απαραίτητη συναγωγή συμπερασμάτων. Ακόμα και στην βοήθεια που χορηγείται για ανάπτυξη πρέπει να ισχύουν οικονομικά κριτήρια τα οποία να είναι γερά θεμελιωμένα στην πραγματικότητα. Πραγματικότητα όμως η οποία αλλάζει διαρκώς. Και αυτές, αυτές τις αλλαγές πρέπει να παρακολουθούν και οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Εγώ προτείνω το EDF να αξιολογεί εάν τα κονδύλια που διαθέτει είναι προσαρμοσμένα στους αναγκαίους δύο στόχους μετανάστευση και προστασία από την τρομοκρατία. Εάν δεν ληφθούν επαρκώ υπόψη αυτοί οι δύο στόχοι, μπορούν, μπορεί να τεθεί σε, κίνδυνο και άλλες πολιτικές Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να διατεθούν σημαντικές πιστώσει λοιπόν, στους στόχους αυτούς, καθώς και στους στόχου που θα ωφελήσουν τις χώρες μέλη. Η ίδια η ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται από την σωστή εξυπηρέτηση των αρχών στις οποίες βασίστηκε η ίδρυσή της προ 70 ετών. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ τις συναδέλφους και τους συναδέλφους για τις εκθέσεις των. Ε, οφείλω να πω, λέει η κυρία Κάρη, ότι υπάρχει πια κάποια μηχανία Αρχίσαμε ήδη να συζητούμε τους προϋπολογισμούς από πέρσι και κάθε φορά διαπιστώνουμε κάποια παράλογα στοιχεία, τα θέτουμε υπόψη του Συμβουλίου και το Συμβουλίο δεν απαντά. Σαν να μας κοροϊδεύει, όχι μόνο εμάς τους ευρωβουλευτές, αλλά και τους πολίτες, το σύνολό τους. Εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε οι θεματοφύλακες των συμφερόντων των πολιτών. Το μόνο που μπορούμε να πούμε σήμερα είναι ότι η Κομισιόν θα πρέπει να είναι απέναντι μας διαφανής και ανοιχτή. Έχουμε θέσει ερωτήσει όμως απαντήσεις δεν λάβαμε. Δεν σημαίνει τίποτε λοιπόν. Ό,τι και αν ζητούμε εμεί, Αυτό δείχνει έλλειψη σεβασμού προς τους πολίτες. Οφείλω να αναγνωρίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχει δουλέψει πολύ και σκληρά. Αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα. εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλό το ποσοστό σφαλμάτων στις ε, διαθέσεις πιστώσεων. Οι ιδέα απαντήσεις της Κομισιόν δείχνουν σαν να θέλει να φορτώσει το βάρος αυτό στις πλάτες άλλων. Δεν μπορούν να διατίθεται τα κονδύλια από τα χρήματα των φορολογουμένων με τόσο πολύ υψηλό σφάλμα. Ναι, ευχαριστώ πολύ και στο συγγνώμη μιλούσατε εκ μέρους της ΓΚΟΕ. Παρακαλώ τον κύριο Σόλτας τώρα για ένα λεπτό. Πράσινη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το ποσοστό σφάλματος στο Ευρωπαϊκό Ταμείο ανάπτυξη είναι υψηλότερο από το ανώτατο επιτροπόμενο όριο για τρίτη συνεχιζόμενη χρονιά δε είναι υψηλό υψηλότερο από το ανώτατο όριο το ποσοστό του σφάλματος. Πιστεύουμε ότι τα περισσότερα σφάλματα θα μπορούσαν να διορθωθούν, να αποφευκθούν, να μειωθούν στο 2% κατά τρόπο ώστε να μπορέσουμε και εμείς να ε, εστιαζόμαστε περισσότερο στις επιτυχίες των ε, προγραμμάτων και των ε, σχεδίων. Η νομότητα, η τήρηση των κανόνων έπρεπε να έχει επιτευχθεί εδώ και πολύ καιρό. Πρέπει να προχωρήσουμε λοιπόν ένα βήμα παραπέρα τώρα και πρέπει να απαιτήσουμε τα έργα να προχωρούν με βάση τους στόχους τους για την εξασφάλιση της ανάπτυξης σε διάφορες περιοχές. Πρέπει να εστιάσουμε στο περιβάλλον, τα κοινωνικά, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος πάλι, παρακαλώ, ένα λεπτό και 30 δεύτερα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο, ο προϋπολογισμός αφορά 150 δισεκατομμύρια τα οποία ανήκουν στο, στα 500 εκατομμύρια κατοίκων. Οπότε θα πρέπει επομένως να ε, είμαστε υπεύθυνοι με διαφάνεια και σχέση με το τι, αν πιάσουν από τα λεφτά. Οπότε χρειάζεται να υπάρχει δημοσιοποίηση όλου του υλικού που έχει σχέση με, με τα ταμεία και πολλές φορές έχουμε κάποιες επενδύσεις ε, μεγάλα έργα ε, όπως το, τη γραμμή των Ρινολιών που κοστίζει πάρα πολύ και δεν ωφελεί. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους ε, διαγωνισμούς που δεν έχουν διαφάνεια σε διάφορες περιφέρειες. Ακριβώς όπως λέει το Ελληνικό Συνέδριο, χρειάζεται διαφάνεια και όσον αφορά τα χρήματα που πάνε στο προσφυγικό. Εκεί υπάρχει η δικαιολογία του κατεπήγοντος, αλλά δεν θα πρέπει να κάνουμε τα λεφτά σε ε, εγκληματίες και σε ε, απαταιώνες. Επίσης και όσον αφορά την προενταξιακή διαδικασία. Θα πρέπει να δοθούν σε όλο τον κόσμο ε, πληροφορίες τι γίνεται με όλα αυτά τα χρήματα που πάνε στην Τουρκία, μια χώρα που καταπατά τα δικαιώματα της διαχείρισης των δικαιωμάτων. Οπότε θα πρέπει να προβληματιστούμε. Επίσης αύριο θα ψηφίσουμε τι γίνεται όσον αφορά τα επιστημονικά δεδομένα τα οποία η, η ΕΦΣΑ η υπηρεσία για τη διατροφική ασφάλεια έχει πει να ξέρουμε κατά πόσον τρώμε δηλητήρια ή όχι. Η Ευρώπη είναι υπέρ της υγείας των ε, πολιτών και η ΕΦΣΑ θα πρέπει να χρησιμοποιεί κάποια δεδομένα τα οποία ε, είναι μετά από έλεγχο των νομοτήμων και από επιστήμονες και μόνο αυτά. Γύρω Σαλίο, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρώτα. Είναι η αρχιτεκτονική πάρα πολύ περίπλοκη και έχουμε τώρα ε, διασπάθηση για διάφορα έργα και δεν υπάρχει διαφάνεια ούτε υπάρχει έλεγχος και έτσι απομακρύνονται οι, τα έθνη και οι λαοί πολλές φορές τα ίδια ε, λάθη γίνονται τη μία χρονιά μετά την άλλη και όλα αυτά τα λάθη ε, τα οποία γίνονται τη μία χρονιά δεν διορθώνται την επομένη οπότε θα πρέπει βέβαια να πούμε μπράβο στο ελληνικό συνέδριο τώρα μπορούν οι βουλευτές να ε, πρέπει καλύτερα. Οπότε το, παραμένουν τα ερωτήματα, τι γίνεται, τι κάνει ο, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τι είναι με τα έξοδα ε, τα εκλογικά, το είπαμε προηγουμένως, οι απαντήσεις που δόθηκαν δεν είναι σαφές. Και είναι περίεργο που τα δύο μεγάλα κόμματα έχουν παραιτηθεί από αυτό το τόσο λεπτό θέμα και θα πρέπει η Όλαφ να επιληφθεί. Το θέμα αυτό μας φέρνει σε αμηχανία και σπηλώνονται έτσι όλα τα θεσμικά όργανα. Κύριος Επιτίδιος έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο ρόλος του Κέντρου Προλήψεως και Ελέγχου Νόσων και η αποστολή που επιτελεί είναι σημαντικά και αξιέπαινα και πρέπει να χρηματοδοτείται οι δραστηριότητε του. Σε μένα όμω γεννούνται τα εξή ερωτήματα. Έχει ενημερώσει κανένα το κέντρο για την απαράδεκτη και τραγική κατάσταση που επικρατεί στον τομέα τη υγεία στην Ελλάδα εξαιτία των απάνθρωπων μέτρων του μνημονίου που έχουν επιβληθεί και από την ευρωπαϊκή ένωση εδώ και έξι χρόνια στον ελληνικό λαό. γνωρίζει κανείς ότι η υγειονομική περίθαλψη στην ελλάδα είναι σχεδόν ανύπαρκτη λόγω του ότι δεν διατίθενται λόγω των μέτρων λιτότητας χρήματα στον ε, υγειονομικό τομέα. γνωρίζετε ότι κάθε εβδομάδα οι διευθυντές των νοσοκομείων σε συνεργασία με τους γιατρούς αποφασίζουν ποιες περιθάλψεις θα περικοπούν. γνωρίζετε ότι δεν υπάρχουν δεν διατίθενται χρήματα για να αγοραστούν φάρμακα που αντιμετωπίζουν τις επικίνδυνες ασθένειες με αποτέλεσμα να πεθαίνουν αβοήθητοι ασθενείς. γνωρίζετε ότι οι προμηθευτές των υγειονομικών υλικών έχουν περιορίσει τις παραδόσεις με αποτέλεσμα οι κλινικές να αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε βασικά υλικά και να υποφέρουν οι ασθενείς. γνωρίζετε ότι έχει περιοριστεί το φαγητό το οποίο δίδεται στα νοσοκομεία. γνωρίζετε ότι όσοι δεν έχουν χρήματα είναι καταδικασμένοι σε θάνατο γνωρίζετε ότι έχει αυξηθεί η θνησιμότητα στην ελλάδα σε πολύ μεγάλο βαθμό. η ελλάδα έχει τις περισσότερες θανάτους από γρήπη από οποιαδήποτε άλλη χώρα της ευρωπαϊκής ενώσεως. τα περισσότερα παιδιά είναι ανεμβολίαστα. έχει αυξηθεί κατακόρυφα η παιδική θνησιμότητα και οι πρόορες γεννήσεις παιδιών που και αυτά πεθαίνουν λόγω του ότι δεν υπάρχει η κατάλληλη περίθαλψη. τι κάνει για όλα αυτά η ευρωπαϊκή ένωση σαν να αποφευθεί η γενοκτονία αυτή των ελλήνων. τίποτε περισσότερο από το να ανέχεται την τουρκία να στέλνει εκατοντάδες λαθρομετανάστες οι οποίοι μεταφέρουν αρρώστιες επικίνδυνες που έχουν εδώ και πολλά χρόνια ξεχαστεί. Ευχαριστώ. Ξεπεράσατε κατά πολύ το χρόνο σας. Τζογόφσκι, μισή λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω την Ίγκε Γκρέσλε και άλλους συναδέλφους Επιτροπής του Ελέγχου του Προπολογισμού για την πάρα πολύ καλή δουλειά που κάνανε για αυτές τις εκθέσεις. Ιδιαίτερα η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού με αργά αλλά σταθερά βήματα καθίσταται μια από τις πιο σεβαστές επιτροπές εδώ στο Κοινοβούλιο, χάρη στη δουλειά της. Και θέλω να επισημάνω τα εξής. Καταρχάς, η υπηρεσία εξωτερικής δράσεως η υπηρεσία της κυρίας Μογκερίνη με άλλα λόγια. Για τη δομή της υπηρεσίας. Είναι υπερβολικά περίπλοκη και άρα αντιπαραγωγική η δομή της. Συστήσαμε περιπτώσεις οποίε χρειάζεται ταχαίως να ληφθούν αποφάσεις, αλλά δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Υπάρχει απουσία ανάλυσης, κάθε διαδικασία προχωρεί με πολύ βραδείς ρυθμούς. Και άλλες διαδικασίες είναι ε, βραδίες, περίπλοκες, πολλές φορές διακόπτονται απότομα πρόσληψη διπλωματών. Έχει αφισβητήσιμα συστήματα, γιατί ορίζονται μόνο από τα παλαιά κράτη-μέλη διπλωμάτες, δεν υπάρχουν από τα νέα κράτη-μέλη. Η λειτουργία των επιτόπου γραφείων επίσης. Επίσης θέλω να επισημάνω ότι υπάρχουν πολλοί που έχουν πει ότι δεν θα συμβάλλουν στη διαδικασία της απαλλαγής. Καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν να δώσει απάντηση και λύση στο μακροχρόνιο αυτό πρόβλημα, ιδιαίτερα σχετικά με τον προπολογισμό του Συμβουλίου, του οποίου η απαλλαγή δεν μπορεί να εξασφαλιστεί γιατί δεν συνεργάζεται. Για ένα λεπτό, ο κύριος Λιμπεράτσκι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, και εσείς κύριε Πρόεδρε του Ελεκτικού Συνεδρίου. Είπε μια ωραία φράση κυρία Τζιαμπάλοβα να μην χρησιμοποιούνται όλα αυτά για πολιτικά παιχνίδια. Δεύτερο, έκθεση Πίπερ, τον οποίο ευχαριστώ για την πολύ θετική συνεργασία του. Είπε ότι η αξία και το νόημα της εργασίας του Ευρωκοινοβουλίου είναι σημαντικά. Η ΔΕ Επίτροπος αναφέρθηκε στη σημασία της μέτρησης με δείκτες και του ποσοστού σφάλματος για τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου το ποσοστό του σφάλματος ήταν τη τάξη του 0,5% και έπεσε στο μισό από πέρσι που ήταν ένα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να ευχαριστήσουμε θερμά τον πρόεδρο Μάρτιν Σούλτς και τον Γενικό Γραμματέα Κλάους Βέλε. Το Κοινοβούλιο πρέπει και να δίνει και το καλό παράδειγμα. Ο κύριος Κερμπράντι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου πρώτα να ευχαριστήσω όλες και όλους τους εισηγητές για τη θαυμάσια εργασία. Τιμώ επίσης την παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βεβαίω και πριν και της ε, Ολλανδικής Προεδρίας. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η απαλλαγή του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διαπιστώνω ότι παρά το γεγονό ότι συζητούμε ακριβώ αυτό το θέμα, ο πρόεδρο μα είναι απόν. Παρόλο δηλαδή που ω κοινοβούλιο καλούμεθα να χορηγήσουμε απαλλαγή στον πρόεδρό μα. Τονίζω και πάλι ότι ο πρόεδρος φαίνεται πως υπάρχει κάποιο πρόβλημα τεχνικό με τις μεταφράσεις. Σημειώνει η πρόεδρο τη συνεδριά. Αποκαταστάθηκε. Καλώ. Συνεχίστε παρακαλώ αγαπητέ κύριε. Να συνεχίσω απλώ ή να ξαναρχίσω. Θα ξαναπώ τότε ότι εκφράζω τη λύπη μου για το γεγονός ότι ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου δεν είναι παρόν, διότι εν τέλει στον πρόεδρο χορηγούμε απαλλαγή. Ελπίζω να του μεταφερθεί το μήνυμα αυτό. Είμαι Ολλανδός. Στον τελευταίο εκλογικό αγώνα ε, διαπίστωσα πόσο ευάλωτοι είμαστε ως θεσμικό όργανο. Ολόκληρος εκείνος ο εκλογικός αγώνας στράφηκε γύρω από την αποζημίωση για δαπάνες των ευρωβουλευτών. Όλα τα υπόλοιπα ήταν δευτερεύοντα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ως Κοινοβούλιο να είμαστε διαφανείς. Στις 16 Απριλίου 2014, προ δύο ετών λοιπόν, είχαμε ψηφίσει ψήφισμα που απίφθινε παράκληση στον Γενικό Γραμματέα να θεσπίσει μια ρύθμιση που να επιτρέπει τον έλεγχο των καταποκοπήν δαπανών μας. Δεν έγινε αυτό τελικά. Τώρα επανέρχεται άλλη τροπολογία με το ίδιο νόημα. Επιθυμώ να παρακαλέσω τους συναδέλφους μου να υπερψηφίσουν, αλλά θα ζητήσω και από την ίδια την Πρόεδρο να φροντίσει ώστε αυτό να γίνει πραγματικότητα. Δέχεστε μια γαλάζια κάρτα, αγαπητέ από τον κύριο Λιμπεράτσκι. Δέχεστε μια γαλάζια κάρτα από τον κύριο Λιμπεράτσκι, κύριε Γερμπράντη. Ορίστε κύριε. Ευχαριστώ. Κύριε Γκερμπράντη, έχω μία ερώτηση. Απευθυνθήκατε στον πρόεδρο Σούλτς σχετικά με τους κορυφαίους υποψηφίους. Ρωτήσατε τον δικό σας τον κύριο Βερχόφστατ που και αυτός ήταν τότε κύριος υποψήφιος αντιμετωπίστηκε με τον ίδιο τρόπο η δική του θέση όπως του Πρόεδρου Σούλτς. Απαντά ο κύριος Κερμπράντη στα αγγλικά αυτή τη φορά. Ίσως επειδή μίλησα Ολλανδικά να μην πέρασε απόλυτα το νόημα. Δεν άσκησα προσωπικά κριτική στον ε, κύριο Σούλτς τον επέκρινα ως πρόεδρο και όχι επειδή υπήρξε βασικός ε, υποψήφιος σπίτσιν candidate αυτό που η ορολογία που πέρασε τότε πιστεύω ότι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου οφείλει να είναι παρόν στην διάρκεια της συζητήσεως για την απαλλαγή που δίνεται στο όργανο χωρίς αυτό να έχει καμία σχέση με το συγκεκριμένο πρόσωπο που ασκεί το αξίωμα αυτό Θεωρώ ότι πρόκειται για μια γενική αρχή. Θεωρώ λοιπόν ότι ο πρόεδρος θα πρέπει να είναι υπεύθυνο και θα πρέπει να είναι παρόν. Δέχεστε μια δεύτερη γαλάζια κάρτα, βεβαίω. Ορίστε κυρία Αγιάλα Σέντερ. Πέστε μου απλώς, σύμφωνα αυτή την αρχή, θα έπρεπε και ο κύριος Γιούνκερ και ο κύριος Τούσκ να παρίστανται. Δεν ήταν να έχει ε, υποβάλει τέτοιο αίτημα, τέτοια τροπολογία. Ελπίζω την επόμενη φορά να το κάνετε. Yes, Mrs. Ayala Sender. I, I do... Ναι, κύριε Ayala Σέντερ, θεωρώ ότι πρόκειται περί σημαντικού θέματος. Επί σειρά ετών επαναλαμβάνω το ίδιο και θεωρώ ότι μια που ε, εδώ εμείς εργαζόμαστε και πάντοτε επικρίνουμε όλους τους άλλους και ιδίως τα άλλα θεσμικά όργανα. Θα πρέπει να ασκούμε και αυτοκριτική και να το κάνουμε συχνά και να κοιτάμε προς τα μέσα, να κοιτάμε εμείς πώς λειτουργούμε. Αλλά συμφωνώ με αυτό που είπατε. Ο κύριος Γιαβόρη το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να μιλήσω για δύο απαλλαγές γιατί είμαι Πρώτα πρώτα για την ΕΦΣΑ. Υπήρχε αυτό το ε, σκάνδαλο για διάφορα διαδικαστικά λάθη και όσον αφορά σύγκρουση συμφερόντων, εμεί θα πρέπει να είμαστε αδαμάντινοι και να μην δώσουμε την απαλλαγή στην ΕΦΣΑ μέχρι ότου αυτό το σκάνδαλο ξεδιαλυθεί. Φωτιστεί τέλο πάντων όσον την απαλλαγή του Κοινοβουλίου. Εμείς λέμε πάντα για διάφορα σκάνδαλα, Lux Leaks, ε, τα Panama Papers και άλλα. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε τι συνέβη και πώς κάποιοι είναι οι υπεύθυνοι. Απ' την άλλη μεριά, απ' την άλλη μεριά οι ευρωβουλευτές ε, δεν διέπονται από διαφάνεια όσον αφορά τα δικά τους έξοδα, όπως και τις ε, γενικές δαπάνες και αποζημίωσή τους και δεν δίνουν λόγο σε κανένα. Θα πρέπει να είμαστε 100% διάφανοι ούτως ώστε να είμαστε αξιόπιστοι και να μην κουράμε το δεύτερο στα άλλα θεσμικά όργανα, αλλά να κάνουμε και αυτοκριτική. Ο κύριος Σάνεμάκης. Θα πρέπει επιτέλους να προβληματιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για το σκοπό τη, το σκοπό της ύπαρξεώ τη και με τον κόσμο. Νομίζω ότι η απαλλαγή είναι μια τέτοια ευκαιρία για να προβληματιστούμε. Πρόκειται για έναν δογματισμό, με μονή θρησκευτικού χαρακτήρα και ε, συνέχεια πληροδοτούμε για περισσότερη Ευρώπη. Αυτό είναι λάθος, αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Είχαμε την κρίση του ευρώ, το μεταναστευτικό. Αυτό είναι τέλεια παράδειγμα. Μα ο κόσμος πια δεν συμφωνεί και εγώ διαμαρτύρομαι εντόνως για αυτή την υπεροψία κατόπιν ε, του πρόσφατου δημοψηφίσματος στις κάτω χώρας για την ευρωπαϊκή πολιτική. Η πρόεδρος κύριε ε, Ντόιτς λεπτό έχετε το λόγο. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο, λέει ο κύριος Ντόιτς. Κυρία Πρόεδρε, Συνάδελφοι, να σας μιλήσω για την έγκριση της απαλλαγής των ε, περιφερειακών υπηρεσιών. πρωτοβουλία συγχαρητήρια στην εισηγήτρια και σε όλους τους σκιώδεις, διότι συνεργάστηκαν πάρα πολύ επικοδομητικά τόσο αφορά τις διάφορες υπηρεσίες η απαλλαγή και η διαχείριση ε, απετέλεσε αντικείμενο ελέγχου από, από την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών για την κάθε υπηρεσία χωριστά και όλες οι υπηρεσίες έλαβαν το πράσινο φως και από το ελεγκτικό συνέδριο εις ε, την διαδικασία των οικονομικών ελέγχων ε, διεκπεριώθηκαν τα όσα εκκρεμούσαν και νομίζω ότι η κατάσταση βελτιώνεται λίγο-λίγο και επίσης για την χρήση 2014 θεωρούμε ότι τα πράγματα πήγαν καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Δεν ε, βρήκαμε λάθη και δεν βρήκαμε λήψεις. Νομίζω ότι ήταν καλή η προσέγγιση. Τα πράγματα ήταν αρκετά έφτακτα. Πριτάνευσε η διαφάνεια στη λειτουργία των υπηρεσιών. Όμως, σε κάποιες υπηρεσίες, όπως είπε και το ελληνικό συνέδριο, υπάρχουν κάποια στοιχεία που επιδέχονται βελτίωση. Όπως στα του ελέγχου της διαχείρισης. Άρα θα πρέπει να βελτιώσουμε την διαφάνεια της λειτουργίας αλλά και την λειτουργία αυτών των υπηρεσιών. Ο, πάντα παρόλα αυτά, εγώ προτείνω να εγκριθεί η απαλλαγή όλων των υπηρεσιών. Ε, ευχαριστώ. Νομίζω ότι έχουμε αυτή την κοινή έγκριση και πρέπει να αποφασίσουμε για όλα μαζί. Πάντως είχαμε κάποιες προστριβές με την εισηγήτρια, αλλά είπαμε για το Clean Sky, το Cesar και, και διάφορες υπηρεσίες ε, τελικά συμφωνήσαμε γιατί πρόκειται για πολύ φιλόδοξες πρωτοβουλίες εκτός την Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί συμμετέχουν και άλλες ε, χώρες. Επίσης όσον αφορά την σύνδεξη ε, είμαστε πρωταγωνιστές ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης έχουμε το Ότομακ που είναι μια μέθοδος αξιοποίησης της θερμοπυρηνικής ενέργειας. Όλα αυτά τεχνολογικά είναι πολύ προχωρημένα, οπότε και πρόκειται για ένα έργο, για ένα πρόγραμμα πάρα πολύ αξιόλογο. Υπάρχουν κάποια προβλήματα και υπάρχει και προπολογισμό που δεν είναι ρεαλιστικός. Όμως, εάν υπάρχει νέα διεύθυνση, νέα διαχείριση, να έχουμε ένα νέο πρόγραμμα δράσης και νέα προσέγγιση. Οπότε θεωρώ ότι όλα αυτά θα τα λάβουμε υπόψη στην επόμενη απαλλαγή. Τόιρε. Ο κύριο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και πρώτα θα ήθελα εξ ονόματο τη ομάδα των φιλελευθέρων να απευθύνω τι ευχαριστίες μα στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την θαυμάσια έκθεση που υπέβαλε. Ευχαριστώ και την κυρία Ματίνα Νταμπάιοβα της δικής μας πολιτικής ομάδας, η συγγήτρια, η οποία έχει δώσει κατευθύνσεις και πληροφορίες που είναι πολύ αναγκαίες. Όλες οι ομάδες μοιράζονται το κοινό αυτό αίτημα της καλύτερης χρήσης των δημοσίων χρημάτων. Υποδομή, ανάπτυξη, παιδεία, κατάρτιση χρειάζονται χρήματα δεν επιτρέπεται να σπαταλώνται άδικα τα χρήματα αυτά. Το ελεγκτικό συνεδρίο έχει δείξει και στο παρελθόν περιπτώσεις όπου δεν είναι σωστά η διάθεση των χρημάτων. Πρωτίστως θέλουμε εδώ έναν προϋπολογισμό που να βασίζεται, που να μετρείται σχετικά με την απόδοσή του. Performance based το λένε στα αγγλικά. Θα χρειαστεί να γίνει αυτό ακόμα συνεπέστερα, η ε, προσπάθεια και ο αγώνας να γίνει ακόμα συνεπέστερη ζητούμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα αιτήματα αυτά και να γίνει σύγχρονο το δημοσιονομικό μας σύστημα. Και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αρχίσουμε και εμείς οι ίδιοι να λαμβάνουμε σοβαρότερα τα όσα λέει το ελεγκτικό συνέδριο, αποδίδοντας και μεγαλύτερη αξία στις έκτακτες και ειδικέ εκθέσεις του που υποβάλλει στις διάφορες ε, επιτροπές. Ε, το ίδιο ισχύει και για τις εκθέσεις που κάνει για την Ελλάδα. Αν χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα αυτά θα καταλήξουμε σε καλύτερη διάθεση των δαπανών. Better spending. Ευχαριστώ. Κύριο Σάρβαμα, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουν επεκταθεί αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής και των άλλων θεσμικών οργάνων και ο προπολογισμό έχει λάβει όλο και μεγαλύτερη σημασία και ο τρόπο διαχείρισή του για τον Ευρωπαϊκό Φορολογούμενο. Αυτό είναι μια γενική παρατήρηση. Γιατί όμω είναι τόσο σημαντική άραγε η απαλλαγή. Είναι σημαντική διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο που εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες και γι' αυτό έχουμε τον κρίσιμο ρόλο να εποπτεύουμε την χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων. Δικός μας είναι ο ρόλος της αύξησης της διαφάνειας, της οικονομικής διαχείρισης και της βελτίωσης της δημοκρατικής λογοδοσίας απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες και πρέπει να γίνουν σεβαστοί οι κοινοί κανόνες. Χρειάζεται να βελτιώσουμε έτσι περαιτέρω την λογοδοσία αυτή, δίνοντας όμως μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα, στην απόδοση και ταυτόχρονα στις απαραίτητες διορθώσεις. Το πιο σημαντικό όμως είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην διαδικασία οφείλει να ενισχυθεί. Αυτό συχνά παραβλέπεται και κατά τη γνώμη μου ο μόνος λόγος είναι ότι δεν του έχει αποδοθεί η θεσμική σημασία που είναι αναγκαία. Όσο η απαλλαγή δεν είναι δεσμευτική, υπονομεύουμε και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά ακόμα χειρότερα την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σάρβαμα. Ακολουθεί η κυρία Κάντενμπαχ για ένα λεπτό μόνο. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, πρώτον ευχαριστώ το ελεγκτικό συνέδριο για την θαυμάσια συνεργασία. Συνεργασία την οποία θα θέλαμε να δούμε και με το Συμβούλιο. Όπως και τα προηγούμενα, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού συνιστά απαλλαγή. Α, να μην δοθεί απαλλαγή εννοώ, αλλά να αναβληθεί. Όπως και σε άλλα προηγούμενα χρόνια, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βασίζεται ή πηγάζει από την έλλειψη συνεργασίας με το Συμβουλίο λόγω της διαφορετικής ερμηνείας των σχετικών διατάξεων. Από χρόνια αρνείται το Συμβούλιο να μας διαθέσει τα έγγραφα τα οποία είναι αναγκαία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην απαλλαγή. Δεν υπάρχει διαφάνεια. Πώς θα δοθούν απαντήσεις στους Ευρωπαίους φορολογούμενους θα πρέπει να αναγνωρίσει το Συμβούλιο το γεγονός ότι ο συνολικός έλεγχος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού θα πρέπει να υπόκειται στις αρμοδιότητες του μόνου πραγματικά εκλεγμένου θεσμικού οργάνου του Κοινοβουλίου. Πρόεδρε, κύριο Σάλη, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχάς να συγχαρέω την συγκητή για την απαλλαγή για τις δύο υπηρεσίες το 2014 η επιλογή ήταν 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ με διαφορετικές χρήσεις απαστολούν 10.000 άτομα. Έχουμε να κάνουμε με μια ε, κατάρτιση προπολογισμού με βάση τις επιδόσεις για τι περισσότερε υπηρεσίε. Ενισχύεται το επίπεδο εκτέλεση του προπολογισμού και η προαγωγή του έργου που προσφέρουν στον πολίτη. Ωστόσο, πρέπει ακόμη να βελτιωθούν οι αρχέ που θα εξασφαλίσουν περισσότερη προσθεμένη αξία και θα εντοπίσουν δυνατότητε για βελτίωση στα μοντέλα των επιδόσεων που μπορεί να αξιοποιηθούν για τις υπηρεσίες. Ε, έτσι λοιπόν πρέπει και τα συμφέροντα των πολιτών αλλά και η διαφάνεια να εξασφαλίζουν ότι θα εξυπηρετείται το συμφέρον του Ευρωπαίου πολίτη οι υπηρεσίε έχουν αναλάβει τα, από την πλευρά του τα κατάλληλα βήματα, ωστόσο υπάρχει ακόμη περιθώριο για βελτίωση σε μια ολιστική προσέγγιση στο δημόσιο τομέα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει οι ευρωπαϊκέ υπηρεσίε και να ενισχύσουν τι προσπάθειέ του για τη βελτίωση των επικοινωνιακών του δραστηριοτήτων, για να ενημερώνονται καλύτερα οι πολίτε για τι ε, ε, δραστηριότητές τους ε, για να είναι ενήμεροι οι πολίτες και πρέπει να αξιοποιηθούν διαφορετικά μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης. Κάποια σημεία χρειάζονται βέβαια βελτίωση, αλλά βλέπουμε σημαντική αλλαγή ε, νοοτροπίας για τις υπηρεσίες χρειάζονται ακόμα καλύτερες δομές επιδόσεων ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Κυρία Γκρέσλε, ένα μισή λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κύριε Αντιπρόεδρε, χαίρομαι που είστε πάλι κοντά μας κύριε Καλτέιρα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την Ολλανδική Προεδρία δε που ε, ήταν παρούσα. Δεν έχουμε συχνά απέναντί μας υπουργού αμήνης. Δεν ξέρω αν σας κάναμε σημαντική εντύπωση. Πάντως να μεταφέρετε στην Υπουργό την εκτίμησή μας. Η ιδέα Ολλανδική Προεδρία είναι ιδιαίτερα ε, ενεργή Τούτη είναι εδώ στη διαδικασία της ε, απαραγής του εδώ τη χρονιά. Νομίζω θα έδινα ένα βραβείο, ιδίως στους διερμηνείς της, ε, του σώματος, οι οποίοι αντιτάχθηκαν στην αύξηση της αποδοτικότητας του έργου τους. Με ειρωνικό τρόπο το λέει αυτό η κυρία ε, και γι' αυτό ενισχύω με τον ε, διάθεσή μου, τον, ε, ενισχύω με τα λόγια μου τον Γενικό Γραμματέα του Σώματος να προχωρήσει στην προσπάθεια αυτή αύξηση αποδοτικότητας. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο θάρρος για αλλαγές, για να προχωρήσουν τα πράγματα προδραστικά. Μιλήσαμε, εδώ άκουσαμε και την Επιτροπή Αναπτύξεως. Υπά, ε, χρειαζόμαστε πληροφορίες. δεν μπορούν να συνεχίσουν τα πράγματα έτσι γιατί αυτό σημαίνει σημαντική μείωση της φήμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αξιοπιστίας της. Ευχαριστώ ένα μισή λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να μπερδεύουν κάποιους τα στοιχεία. Είναι όμως φυσιολογικό το επίπεδο του σφάλματος στο τέλος μιας ε, περίοδου εκτέλεσης να αυξάνεται. Χωρίς όμως να δείχνουμε περιβολική καχυποψία, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι την ώρα της απαλλαγής διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν όργανα με τα οποία συνεργαζόμαστε καλά και θα ήθελα να ζητήσω στην επόμενη απαλλαγή ιδιαίτερα να δώσουμε έμφαση στις εκρεμείς πληρωμές, στους ανεξόφλητους λογαριασμούς. Μόνο έτσι μπορούμε να φτάσουμε στο στόχο του, ε, της Ευρώπης 2020. Μόνο έτσι μπορούμε να υπηρετήσουμε τη δημοκρατία και αυτό πρέπει να καταστεί ορατό για τον κάθε πολίτη έξω από το κοινοβούλιο. Να δει δηλαδή ότι τα ευρωπαϊκά μέσα τα αξιοποιούμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγχονται και αν έχουν σωστά απορροφή στα κονδύλια να εξασφαλίζουν περισσότερη χρηματοδότηση. Η Βουλγαρία ιδιαίτερα, με ιδιαίτερη προσοχή ε, χρησιμοποιεί την ε, ε, νομοθεσία για τις δημόσιες προμήθειες και μπόρεσε να αξιοποιήσει με πολύ ικανοποιητικό τρόπο τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση και στο θέμα, των, συγγνώμη, στον κατάλογο των ομιλητών εκ μέρους των ομάδων και τώρα θα δώσουμε το λόγο στη δικασία Καρστιάη με την κυρία Σόιτροβα πρώτη. Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ζητώ το λόγο για την απαλλαγή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014 για να υποστηρίξω το βραβείο ταινιών Λουξ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επιστήσω την προσοχή στον κίνδυνο που το απειλεί. Οι δαπάνε του 2014 για το βραβείο αυτό ε, μειώθηκαν στο 391.000 ευρώ και αυτό ε, μείωσε τις δυνατότητες και υποτιτλισμού και ε, προβολής της ταινία. Αυξήθηκε για το 2015 στα 193.000 ευρώ ο προϋπολογισμός ε, για την προβολή των ταινιών αυτών σε 28 χώρες και 41.000 θεατές. Οι δαπάνες λοιπόν είχαν μια μικρή διαφορά στα 500 περίπου στα 550 ευρώ με μια πολύ σημαντική δραστηριότητα όμως για την υποστήριξη των ε, ευρωπαϊκών αξιών ο κ. Μαριάς ο ΕΝΙΣΑ αποτελεί το μοναδικό αποκεντρωμένο οργανισμό της ευρωπαϊκής ένωσης που βρίσκεται στην ελλάδα η οποία έχει δαπανίσει εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της λειτουργίας του οργανισμού. κυρία γεωργίευα ο ΕΝΙΣΑ διαθέτει υπερσύγχρονα γραφεία τεσσεράμισι τετραγωνικών μέτρων στο ηράκλειο της κρήτης. στα γραφεία αυτά όμως δυστυχώς απασχολούνται μόνο δέκα άνθρωποι αφού το επιχειρησιακό κέντρο του οργανισμού μεταφέρθηκε στην αθήνα παρά το γεγονό ότι οι ελληνικές αρχές υλοποίησαν όλες τις δεσμεύσει που είχαν αναλάβει για τη λειτουργία του ενίσα στο ηράκλειο. δυστυχώς στις 16 μαρτίου η επιτροπή προπολογισμού του κοινοβουλίου στήριξε τις μεθοδεύσει της διοίκηση του ενίσα και άνοιξε ουσιαστικά το δρόμο για απαξίωση του οργανισμού στο ηράκλειο. Τελικό στόχο τη μεθόδευση τη ηγεσία του ενίσα είναι η μεταφορά τη έδρα στι βρυξέλλες από το 2012, χιλιάδες δώδεκα ως βουλευτής ηρακλείου δίνω αγώνα με τις τοπικές αρχές για να σταματήσουν οι μεθοδεύσεις της ηγεσίας του ενίσα η οποία ήρθε την περασμένη εβδομάδα εδώ στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο με αλαζονικό ύφος και ηρωνευόταν τους ευρωβουλευτές. κυρία γεωργίευα παρακαλώ να εξετάσετε το θέμα του ενίσα σοβαρά. σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εσάς ε, κύριε Πρόεδρε του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Μιλούμε για την απαλλαγή 53 συνολικών ε, οργανισμών και άλλων φορέων. Από τις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο ευχαριστούμε ιδιαίτερος, διαπιστώνουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά αδύναμα σημεία στις δημοσιονομικές βοήθειες που δίνονται και αυτό οφείλεται στην, στους ελληματικούς ελέγχους. Επομένως, σε διαδικασίες, σε μείωση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. Για πέντε οργανισμούς σημειώθηκαν, ε, διαπιστώθηκαν σημαντικά σφάλματα. μεταξύ αυτών ο Frontex, η Ευρωπαϊκή Αρχή Περιβάλλοντος, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την πρόληψη των ασθενειών. και μιλούμε για ε, δαπάνες της τάξης των 47 εκατομμυρίων ευρώ. Εκεί δεν έχουν αναζητηθεί επαρκώς, για παράδειγμα, πόροι οι πηγές ιδιωτικής χρηματοδότησης. Γι' αυτό εγώ ζητώ τροποποίηση των κανονισμών της δημοσιονομικής βοήθειας. Ο κύριος Πόλτσακ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρώτα-πρώτα, χαίρομαι ε, που με τις κοινωνικές επιτροπές αλλά και τους εισηγητές απέκτησε ενδιαφέρον ε, αυτή η υπόθεση και εκτιμώ πάρα πολύ την εισηγητρία. Κοιτάξτε, θέλω να πω τι γίνεται με όλε αυτέ τι εκκρεμούσε πληρωμέ, τα είπαμε και τα ξαναείπαμε. Νομίζω ότι αυτή η καθυστέρηση για τα πολιετή ε, ταμεία και για την πολιτική συνοχή είναι κάτι ε, το οποίο επιδέχεται κριτική. Ε, αυτού του είδους η καθυστέρηση των πληρωμών ε, αφορά κάποιους αποδέκτες, κάποιους δικαιούχους που έχουν θεμητές προσδοκίες δεν θα έπρεπε να γίνεται κάτι τέτοιο. Και όσον αφορά την Περιφερειακή Επιτροπή τα έχουμε πει και επικρίνει επανειλημμένα. Ε, πάρα πολύ σωστά αυτά που λέει η σχετική έκθεση και θα πρέπει να προσέξουμε και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις αλλά και τα πολιτικά προγράμματα. Ε, Είναι πολύ σημαντικό το Κοινοβούλιο να υποπτεύει τον λογαριασμό και το, τον προπολογισμό και να Προσέγγιου ούτως ώστε να πιάνουν τόπο τα χρήματα και τα προγράμματα, κάτι για τα πιλωτικά προγράμματα. πρώτοι για έναν τομέα που θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα, ιδίω όσον αφορά τα σχέδια με το COP21. Και ο κύριος ε, Γιάννη και είπε ότι θα πρέπει να είμαστε πιο πρωτοπόροι για την καινοτομία, για τα πιλωτικά προγράμματα και τα σχετικά. Επίσης, θα ήθελα να σταθώ δύο λίγο σε κάτι άλλο το οποίο δεν το έχουν περιλάβει στην ημερική διάταξη τους ιδίους πόρους. Τα συζητήσαμε στην τελευταία εντολή, αλλά δεν τα συζητήσαμε τώρα. Σήμερα τα κρατημέλη να αυξήσουν την συμβολή τους. Υπάρχει όλο ένα και περισσότερη συζήτηση και άρα θα πρέπει στη χρηματοδότηση να περιλαμβάνονται οι ίδιοι πόροι. Ευχαριστώ. Φτάσαμε τώρα στο τέλο ε, ε, ε, τη διαδικασία διαδικασίας Ο κύριο Καλτέρα έχει το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τα καλά σας λόγια, για τη δουλειά του ελεγκτικού συνεδρίου. Είναι πολύ ενθαρρυντικά για μας. Καλωσορίζουμε όλες τις συστάσεις για τη μελλοντική ελεγκτική δουλειά για τις διάφορες εκθέσεις απαλλαγής. Ιδιαίτερα σημειώνω το αίτημα να συνεχίσει το ελεγκτικό συνέδριο να αναπτύσσει μια διαδικασία βελτίωσης της ε, εξέτασης απαλλαγής της Επιτροπής για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020. Σημειώνουμε τις ε, παρατηρήσεις για τις συμπράξεις και την κοινή ενημέρωση και την βελτίωση της ενημέρωσης για σύσταση που αφορά τη διαδικασία απαλλαγή που προτείνει που ισχυρίζεται ότι είναι μεθοδολογικό το πρόβλημα στο πόσο του σφάλματος και πρέπει να επιληθεί μεταξύ ελεγκτικού συνεδρίου και επιτροπής, δεν νομίζω ότι μπορεί να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε. Αυτό που έχουμε να αντιμετωπίζουμε είναι να ε, αντιμετωπίσουμε τη ρίζα του προβλήματος. και είναι ευπρόσδεκτες οι δηλώσεις της κυρίας Τζορτζίεβα της ε, Επιτρόπου για τον κίνδυνο. Αυτός ο οποίος συντάσσει την νομοθεσία και αυτός που συμφωνεί ως προς τη χρηματοδότηση ενός σχεδίου, ενός προγράμματος πρέπει και να ορίσει μέχρι ποιο επίπεδο κινδύνου μπορεί να φτάσει. Μη στάτε από τους ελεγκτές του προϋπολογισμού να το πράξουν αυτό. Ο ελεγκτής απλώς θα επαληθεύσει εάν υπάρχει υλικό επίπεδο σφάλματος. Καταγράφω λοιπόν την πρόταση, αλλά εάν θεωρείτε πως πρόκειται για μία λύση, δηλαδή για θεώρηση του προβλήματος των σφαλμάτων ως μεθοδολογικού ζητήματος που μεθοδολογικά πρέπει να αντιμετωπιστεί, δεν νομίζω ότι οδηγούμαστε σε λύση. Μια νέα προσέγγιση των σφαρματων ως θα πρέπει να χρειάζεται ως προς τις δαπάνες και τις επενδύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μέλλον. Πρόκειται για μια πρόκληση κοινή σε όλα τα θεσμικά ε, όργανα Ήδη έχουμε ξεκινήσει να προσπαθούμε προ την κατεύθυνση αυτή. Τρει γραμμέ δράση, τι οποίε μπορεί να συμβάλλει το Ελεγκτικό Συνέδριο. Καλωσορίζουμε και την πρόσκληση του Συμβουλίου να συμβάλλουμε στο, στη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση του του δημοσιονομικού πλαισίου. Καλωσορίζουμε επίση την ευκαιρία να προσφέρουμε απόψει και γνώμε σε σχέση με την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού, που είναι και μια πολύ σημαντική στιγμή και θα μα επιτρέψει να ε, χαράξουμε το δρόμο για το μέλλον, αλλά και θα πρέπει να επικεντρωθούμε και στους ιδίους πόρους. Και σε αυτό με την ιδιότητά μας ως ελεγκτών συμβάλλουμε ήδη. Σας βεβαιώ λοιπόν ότι από πλευράς μας θέλουμε και εμείς να συμβάλλουμε σε αυτόν τον διοργανικό διάλογο, ο οποίος θα πρέπει να μεταφραστεί όμως σε συγκεκριμένη δράση, σε απτή δράση. ώστε στο μέλλον να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, καλύτερη δημοσιονομική διαχείριση και λογοδοσία για κάθε Ευρωπαίο πολίτη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Καλντέρα και τώρα το λόγο θα λάβει η Επίτροπος. Κυρία Γεωργίευα έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη γιατί χρησιμοποίησα και δύο λεπτά πριν στην αρχική μου ομιλία. Θα έρθω σε τρία ειδικότερα θέματα. Πρώτα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τις συζητήσεις που, για τη συζήτηση μάλλον που έγινε σήμερα με διάφορες τοποθετήσεις αλλά και για τη συγκεκριμένη αίτηση που μου έγινε να προσέξω. Σας διαβεβαιώ ότι θα εξετάσουμε πολύ προσεκτικά και θα απαντήσουμε στα σχόλια που μας έγιναν σήμερα. Εξάλλου, σημαντικό είναι να σας τονίσω ότι εγκύπτουμε τώρα και στα ψηφίσματα για το follow-up μετά από την απαλλαγή και επίσης και για φέτος. Ακούγοντας τα σχόλια που έγιναν, λέγω ότι βεβαίως πρέπει να συνεχίσουμε να εξετάζουμε προληπτικές δράσεις, διορθωτικές δράσεις στην πλευρά των σφαλμάτων. Είναι πολύ σημαντικό. Το έργο αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με το ελεγκτικό συνέδριο με στόχο να εντάξουμε καλύτερα στις προσπαθειές μας τα διδάγματα που λαμβάνουμε και από τις εκθέσεις τους αλλά και από τη δική μας εργασία. Ο πρόεδρος Καλντέιρα δεν θα δείξει κατανόηση αν δεν το τονίσω. Θα συνεχίσουμε δηλαδή να εξετάζουμε το θέμα του πολιετούς χαρακτήρα των προγραμμάτων μας. Θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε για ένα μακρότερο χρονικό διάστημα να επιτύχουμε τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τα ασφάλματα. Ταυτόχρονα όμως είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες σε όλες και όλους εκείνους που μίλησαν για αναγνώριση των πραγμάτων που τα καταφέρνουμε καλά εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βεβαίως και το ελεγκτικό συνέδριο το αναγνωρίζει στις εκθέσεις του. Δηλαδή μπορούμε να βασιστούμε και στα όσα καταφέρνουμε καλά, ιδίως στην πλευρά της πολιτικής και να μπορέσουμε να πολλαπλασιάσουμε τις καλές πρακτικές έτσι ώστε οι καλές πρακτικές, μάλιστα ακόμα καλύτερα, οι βέλτιστες πρακτικές να γίνουν οι συνήθεις πρακτικοί. Η δέσμευσή μας να συνεργαστούμε και με εσά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με το Ελεγκτικό Συνέδριο και με το Συμβούλιο είναι απόλυτα ε, σίγουροι να βασίζεστε και σε μένα και στο προσωπικό μου θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η διαδικασία αυτή να μην μείνει μια εφάπαξ μόνο περίπτωση αλλά να συνεχιστεί διαρκώς. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Το λόγο τώρα λαμβάνουν οι εισηγητές και πρώτα η κυρία Γκαμπάγιοβα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας καλησπέζω για τρίτη φορά απόψε. Ευχαριστώ για όλες τις θετικές σας ε, παρατηρήσεις και την υποστήριξή σας και πιστεύω ότι αύριο την ώρα της ψηφοφορίας ε, θα πετύχει το εγχείρημά μου σε σχέση με αυτή την τέτοια της απαλλαγής και ευχαριστώ της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού. Ε, όλοι πάρα πολύ δυναμικά με βοήθησαν σε όλη τη διαδρομή και επίσης να συγχαρώ όλους τους συνεισηγητές της ε, Επιτροπής μας για ε, την έκθεση για τις ε, απαλλαγές. Ευχαριστώ και τους εκπροσώπους των άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Συνεργαστούμε πολύ καλά. Να ευχαριστήσω βέβαια για την κυρία Γεωργιέβα, την Επίτροπο, αλλά και τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Και η φιλοδοξία μου ήταν να έχουμε διαφάνεια και να έχουμε μια προσέγγιση των ε, προγραμμάτων και να έχουμε μια σφαιρική προσέγγιση υπό όφελο των Ευρωπαίων και όλα αυτά νομίζω ότι θα αντικατορίζονται στο κείμενο επί το οποίο θα ψηφίσουμε αύριο. Ελπίζω αυτή η προσέγγιση να υιοθετηθεί και για την ε, διαδικασία απαλλαγή του 2015 που θα αρχίσει ε, σε λίγους μήνες. Οπότε ελπίζω ότι οι προτάσεις για τη δημοσιονομική πολιτική θα αγκαλιαστούν και από την επόμενη Δημοσιονομική ε, Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού αλλά και από τι άλλε δημοτικέ επιτροπέ και εν κατακλείδη νομίζω ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί ο διάλογο μεταξύ θεσμικών οργάνων και να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη και να έχουμε κάποιες ομάδες εργασίας που να ε, εποπτεύουν στα αποτελέσματα των προσπαθειών μας και ε, θα πρέπει να κάνουμε κάτι σαν το ευρωπαϊκό εξάμεινο που ήταν συνεχής η συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων επί τη βάση συγκεκριμένου ε, χρονοδιαγράμματος. Έτσι θα μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τον ποσοστό φάλματος και θα αποφύγουμε τα σκάνδαλα που υπονομεύουν την αξιοπιστία μας. Ελπίζω ότι η προσέγγιση μου για την άσκηση του 2014 θα βοηθήσει από βάθους καρδίας. Επίσης, συμφωνώ όλους όσους έλαβαν ε, μέρος από όλα τα θεσμικά όργανα για αυτήν την διαδικασία. Όλοι ήταν πάρα πολύ υπεύθυνοι. Η πρόεδρος Σμιτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εσείς κύριε Επίτροπε και εσείς κύριε Πρόεδρε. Πολλά λέχθηκαν σήμερα. Μια σύντομη αντίδραση ως εισηγήτρια δεν θέλουμε, έχω να πω το εξής, δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε μόνο τα προβλήματα των ε, μεταναστών. Θέλουμε να μπορούμε να αντιδρούμε ταχαίως σε όλες τις προκλήσεις. Και δεν πρόκειται μόνον, και παρακαλώ προσέξτε τι λέω, δεν πρόκειται να ταχθούμε προστατευτικά απέναντι σε πράγματα τα οποία δεν έχουν αποδώσει, ούτε σε πρόσωπα. Χρήματα της αναπτυξιακής βοήθειας, χρήματα τα οποία διαθέτουν οι φορολογούμενοι, θέλουμε να διατεθούν με τρόπο κατάλληλο, επαρκή και χρήσιμο. Ευχαριστώ για την ε, συνεργασία και ελπίζω αύριο να υποστηρίξετε την έκθεσή μου. Ευχαριστώ ε, κυρία Ευρωβουλευτά και ευχαριστώ που τηρήσατε το χρονικό σας όριο. Ο κύριος Πίπερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις προτάσεις και τις επικρίσεις σχετικές με την ε, έκθεσή μου. Διαπιστώνω καταρχάς ότι υπάρχει σε σχέση με τις υπηρεσίες των οδηγών και την ε, όλο και πιο εσωτερική οργάνωση των διαφορών υπηρεσιών για τους βουλευτές μια αλφα δυσκολία σε επίπεδο διοίκησης. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις στις οποίες αναφέρομαι και που δίνουν ε, νομίζω πολύ θετικό φως για την ε, διοίκηση, για την ανεξαρτησία και την εκτέλεση της εντολής. Χαίρομαι και ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη που μου προσέφεραν οι συνάδελφοι. Προς τους φιλελευθέρους και τον κύριο Γκερμπράντη συγκεκριμένα θα ήθελα να πω το εξή ότι η έκθεση απαλλαγής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εάν στηριχθεί κατά την προεκλογική εκστρατεία στην ε, καταποκοπή αποζημίωση εξόδων χωρίς τίποτε περισσότερο, αυτό νομίζω καθίσταται ένδειξη πνευματικής φτώχειας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επιχειρημάτων. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω θα ήταν καλό να έχουμε πιο πολύ ε, ουσιαστικά επιχειρήματα. Τον επικρίνεται επίση τον κύριο Σούλτ, επειδή είναι παρόν εδώ. Και μου απευθύνεται και εμένα ερώτηση όταν δεν είσαστε εσεί ο ίδιο εδώ. Κύριε Κερμπράντε, παρακαλώ. Τουλάχιστον να έχετε το θάρρο να μείνετε στην αίθουσα για να ακούσετε και την απάντηση. Τελευταία παρατήρηση για την κυρία Γκρέσλε που το επεσήμανε Είχαμε πολλά ζητήματα, το κόστος των διερμηνέων, τα, την κεντρική πολιτική, τα διάφορα προνόμια. Κάθε ε, ομάδα εδώ ε, έχει ένα πολύ ισχυρό λόμπι, λέει ναι κάντε οικονομίες αλλά όχι στη δική μου την περίπτωση. Όχι στη δική μου την περίπτωση. Αν λοιπόν υποχωρήσουμε εναντί αυτού, ω Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού δεν καταφέρουμε τίποτα. Για άλλη μια φορά λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω θερμά εκείνου οι οποίοι ε, έδειξαν αιμονή σε μια κοινή θέση, έκαναν προσπάθειες με θετικό πνεύμα και κατάφεραν να βελτιωθούν τα πράγματα. Είναι θέματα εθνικά, ευρωπαϊκά, είναι συμφέροντα των εργαζομένων, είναι όλα αυτά που εκφράζει η απαλλαγή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γι' αυτό πρέπει να την προωθήσουμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τσανέσης και το λόγο. Παρακαλώ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κυρία Γεωργίευα, κύριε Καλτέιρα, αγαπητή Ολλανδική Προεδρία, θα μιλήσω τώρα πολωνικά, πριν μίλησα αγγλικά. Θα μιλήσω για τρία λεπτά για να πω ότι η συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου και κυρίως της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού και του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Λουξεμβούργου είναι πολύ πολύ καλύτερη από ό,τι πριν από 6-7 χρόνια που μπορώ εγώ να θυμάμαι. Εν τέλει βλέπουμε ότι είμαστε στην ίδια, στην ίδια ομάδα, ανήκουμε στην ομάδα των ελεγκτών της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και απευθύνουμε ένα καλό θετικό μήνυμα προς τον Ευρωπαίο φορολογούμενο και κάθε άλλον που θέλει να εκτελείται σωστά ο προϋπολογισμός, να δαπανώνται σωστά τα κονδύλια. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο που θέλω να γύρω είναι ότι πρέπει απερίφραστα να μιλούμε και για τα θέματα της διπλωματικής μας υπηρεσίας, της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης και να ορίσουμε ότι χρειάζεται ε, να επιβληθούν και γεωγραφικές ποσοστώσεις, ποσοστώσεις προελεύσεως, γιατί βλέπουμε ότι από 128 επικεφαλής αντιπροσωπιών στις αντιπροσωπείες Ευρωπαϊκής Ένωσης. 60 προέρχονται από τα κράτη-μέλη και από αυτούς τους 60 μόνο 20 από τα λεγόμενα νέα κράτη-μέλη. Είναι προφανή η δυσαναλογία. Με την αναλογία πληθυσμού η χώρα μου, η Πολωνία, θα έπρεπε να έχει 12 πρεσβευτές Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει μόνο 4. Είναι δυσανάλογο λοιπόν αυτό το γεγονό και δεν αφορά μόνο την Πολωνία, αλλά και άλλα λεγόμενα νέα κράτη-μέλη. Όμω η συζήτηση δεν αφορά μόνο την υπηρεσία εξωτερική ε, δράση. Έχουμε αντίστοιχε καταστάσει και σε άλλα θεσμικά όργανα. Το Κοινοβούλιο δεν έχει τόσο καλές, δεν έχει τόσο κακές επιδόσεις. Το Συμβούλιο όμως είναι το χειρότερο. Και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όταν μιλούμε για το Συμβούλιο λοιπόν έχουμε την εντύπωση ότι χρόνο με το χρόνο βλέπουμε να διαδραματίζεται η ίδια, ε, το ίδιο θεατρικό έργο, το ίδιο έργο. Διαμαρτυρόμαστε εμεί για το Συμβούλιο, εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας γιατί δεν ε, εκφράζει την πολιτική βούληση του Συμβούλιο, λέμε τα ίδια και τα ίδια και βεβαίω έχουμε δίκαιο, γιατί πάντα έχουμε δίκαιο. Μιλάμε λοιπόν, απαντήσεις δεν παίρνουμε και προφανώς είναι προβληματική επικοινωνία. Έχει έρθει η ώρα λοιπόν να ακολουθήσουμε πιο, πιο σκληρή στάση αφού δεν συνεργάζονται τα δύο όργανα λόγω απουσίας βούλησης του Συμβουλίου για συνεργασία. Ευχαριστώ. Δίστησαν δύο λεπτά. Παρακαλώ. Øh, lang debat, men jeg synes, den øh, har bragt øh, os fremad. Jeg gerne både for Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο σκιώδεις συζητητές γιατί με βοήθησαν σημαντικά κατά τη σύνταξη της έκθεσης. Επίσης να ευχαριστήσω την συγκέντρια για την γενική απαλλαγή. Νομίζω ότι ε, όλα τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Θα πρέπει να ε, ασκούμε έναν αυστηρό έλεγχο ε, όσον αφορά τον κοινωνικό προπολογισμό, δεν θα πρέπει να δεχόμαστε τη διασπάθηση, θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα σημεία όπου υπάρχουν προβλήματα. Αξίζει επίση να ισχύουν τα ίδια για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως και για τα άλλα θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ για τη συζήτηση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ελληνικό Συνέδριο για όλη του την βοήθεια για τη στήριξη τη έκθεση. Και με μπορεί θα γίνει η ψηφοφορία και θα ακολουθήσουμε την γραμμή που αποφασίστηκε η Πρόεδρος. Και τώρα ολοκληρώνεται ο κατάλογος των αγορητών εισηγητών.